Γεια σας. Συνεχίζεται η συνεδρίαση. Είμαστε στο σημείο 11 στη σημερινή διάταξη. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω θερμά. Και το συνάδελφο Βιώτη. Ε, και ε, χαιρόμαστε που σας βλέπουμε για να μας ενημερώσετε για τις προτεραιότητες και το κέντρο βάρους, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε ποιες θα είναι και δικές μας. Ο δικός μας, ο δικός μας ε, εισηγητής για την απαλλαγή δεν έχει έρθει ακόμα, αλλά ελπίζω να τα ακούσει στη συνέχεια. Σημειώνεται 11 λοιπόν, για ειδικό Προπολογισμό της Ένωσης. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστούμε την ε, Επιτροπή σας. Ευχαριστώ ε, που μου δίνετε αυτόν τον ε, χρόνο. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Θα κάνω βέβαια κάποιες γενικές παρατηρήσεις μεθοδολογικής υφής αλλά και επί της ουσίας όσον αφορά το θέμα το οποίο αφορά την Επιτροπή σας που ελέγχει τις ε, δαπάνες κατά κάποιο τρόπο. Ε, γιατί προηγουμένως ήμουνα στην Επιτροπή Πολιτισμού και χρειάστηκε ε, να αναφερθώ σε άλλα στοιχεία. Όσον αφορά την μεθοδολογία. Είμαι άλλωστε και με δύο συναδέλφους που προέρχονται από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Ε, δεν είναι εύκολη η διαδικασία. Εγώ προτίθεμαι στις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες να εργαστώ έτσι ώστε ε, ε, γύρω από τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μπορέσω να δημιουργήσω την μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία και την μεγαλύτερη δυνατή συμμαχία ή συνασπισμό συνεργαζόμενος με όλες τις πολιτικές πολιτικές ομάδες ε, του Κοινοβουλίου αλλά και με τις επιπές. Γι' αυτό λοιπόν θα προσπαθήσω όσο γίνεται να βρω την μέγιστη δυνατή συνένεση ε, γύρω από τη θέση μας γιατί είμαι πεπισμένος όταν θα γίνει ε, αυτή η δύσκολη στιγμή της διαβούλευσης με το Συμβούλιο θα πρέπει να υπάρχει ένας εισηγητής όπως έγινε και με τους συναδέλφους των προηγουμένων χρόνων ένας εισηγητής έλεγα που θα έχει όσο γίνεται μεγαλύτερη συνένεση από πλευράς του Κοινοβουλίου έτσι ώστε η διαπραγματευτική του θέση να είναι ε, όσο γίνεται πιο καλή. Η δεύτερη σκέψη που θέλω να κάνω εδώ ενώπιόν σας ε, όσον αφορά πάντα την μεθοδολογία αφορά πρώτον το ρόλο του Συμβουλίου διότι γνωρίζετε ε, ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης είναι άκαμπτος. Είναι δύσκολο δηλαδή να ε, βρει κανεί περιθώριο ελιγμού, ε, καθώς επίσης και να εισάγει και κάποια στοιχεία καινοτομία για να μην πω έτσι εκμοντερνισμού. Δεύτερο στοιχείο είναι ότι πολύ συχνά βρισκό, έχουμε απέναντί μας ένα συμβούλιο το οποίο είναι ακόμα πιο άκαμπτο όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Και επομένως θα πρέπει να έχουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη πολιτική διαπραγματευτική ικανότητα οι προτεραιότητες τις οποίες ε, εγώ έχω καθορίσει και τις οποίες ε, εσείς ε, γνωρίζετε λόγω των guidelines των κατευθυντηρίων γραμμών που ψηφίσαμε τον Μάρτιο δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες καινοτομίε, επικεντρώνονται όμως σε δύο ουσιαστικά στοιχεία που είναι αφενός η αύξηση, δηλαδή παρά τα νέα αιτήματα των νέων προγραμμάτων, νέων επενδύσεων προς του Κοινωνικού Συμβουλίου να ε, ε, διατηρηθούν τα προγράμματα ε, τα οποία αφορούν τους πολίτες, που αφορούν τα ερευνητικά κέντρα, που αφορούν τα πανεπιστήμια, που αφορούν δηλαδή όλες τις προσδοκίες των πολιτών και που μέχρι στιγμής έχουμε δει ότι έχουν δημιουργηθεί, έχουν χρησιμοποιηθεί συγγνώμη, αποτελεσματικά και με τρόπο πλέον επωφελή. Και βεβαίως θα πρέπει όσο γίνεται να υπογραμμίζουμε την κοινωνική πτυχή και το κοινωνικό πρόσωπο της Ευρώπης. Ε, επανειλημμένα έχω συζητήσει για το θέμα αυτό και με άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές ε, με την Επιτροπή ας πούμε ΕΜΠΛ εργασίας. Ε, εκεί υπάρχουν πολλές ε, εκπεφρασμένες προσδοκίες για την κοινωνική υπόσταση της Ευρώπης. Εκεί εντάσσονται οι μεγάλες προτεραιότητες. Επίσης υπάρχουν τα νέα προγράμματα και επ' αυτών θα ήθελα κυρίως να αναφερθώ στο νέο πρόγραμμα για την έρευνα όσον αφορά τον τομέα της άμυνας. Πρόκειται για ένα σημαντικό πρόγραμμα, ε, στο οποίο εγώ πιστεύω πάρα πολύ. Οι επενδύσεις στο νέο πρόγραμμα άμυνας όμως δεν θα πρέπει να σημάνουν ή να προκαλέσουν περικοπές σε άλλα προγράμματα, γιατί και αυτά είναι εξίσου σημαντικά. Και πιστεύω και εδώ μπαίνουμε στα χωράφια της Κοντ περισσότερο, ότι θα πρέπει να συζητήσουμε πολύ το θέμα της εισαγγελία. Δεν έχει ευρωπαϊκή εισαγγελία, δεν έχει ακόμα θεσπιστεί αλλά θα πρέπει επισήμω, αλλά θα πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί από το 2019. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ε, τον προϋπολογισμό του 2019, με ποιο τρόπο θα ενταχθεί εκεί πώς μπορούν να προκύψουν τροποποιήσεις έτσι ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες επενδύσεις και τα απαραίτητα, ε, οι απαραίτητοι πόροι για την ε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορούν να προκύψουν από την Eurojust, από την Olaf ε, και όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους, προσωπικό κτλ. Πάντως εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι η Εισαγγελία θα πρέπει να έχει την δυνατότητα την επόμενη χρονιά να μπορέσει να αρχίσει να λειτουργεί. Το τελευταίο που θέλω να πω, ξέρω ότι η Επιτροπή Κοντ ε, ε, δίνει μεγάλη σημασία στο πρόγραμμα Global Europe, ακριβώς λόγω του ότι ε, ε, και λόγω της απόφασης του δικαστηρίου έχουν ε, απομονωθεί κάποια και διαπιστωθεί κάποιες δυσκολίες και επομένως κυρίως όσον αφορά την Τουρκία και την Αλβανία θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία. Βεβαίως περιμένω και τις δικές σας σκέψεις και τις δικές σας παρατηρήσεις και σχόλια και όσον αφορά την σημερινή μας συζήτηση, αυτή που θα κάνουμε τώρα, αλλά ε, και όσον αφορά ε, την γνωμοδότηση την οποία ε, ενδεχομένω θα μου στείλετε μέσα στις επόμενες εβδομάδες λαμβάνοντα υπόψη ότι εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να κλείσει ε, η σχέση ανάμεσα στον υποφαινόμενο και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές τόσο γρήγορα και οπωσδήποτε θα πρέπει να διατηρηθεί μέχρι τη στιγμή που θα προχωρήσουμε σε διαβούλευση για το θέμα αυτό του προϋπολογισμού. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω ειλικρινά να σας ευχαριστήσω και για τη δική σας ειλικρίνεια. Υποθέτω τις ειλικρινές. Εμείς δυσκολευόμαστε, γιατί είμαστε η Επιτροπή που εφαρμόζει, που υλοποιεί τον προϋπολογισμό. Όλοι επικεντρώνονται στα ποσά στην αρχή και κανένας δεν ενδιαφέρεται για το τελικό αποτέλεσμα. Έχουμε μια παράκληση, πάγια, εδώ ε, και χρόνια, αλλά ανέκαθεν κάνουμε μια τρύπα στο νερό λόγω του Συμβουλίου. Ο προϋπολογισμός για την Εποπτική Επιτροπή της Όλαφ έχει παγώσει εδώ και χρόνια 100.000 ευρώ, ανεξαρτήτως αλλαγή του κόστους. Προσπαθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια να το αυξήσουμε κατά 20% και είναι σχετικά γελίο το ποσό και ποτέ δεν το καταφέραμε. Και συνήθως έχει προσκρούσει αυτό στην αντίσταση του Συμβουλίου. Παρακαλώ ε, να το ζητήσετε κι εσείς μαζί μας και στα τελευταία λεπτά της αντιπαράθεσης θα πρέπει να το πείτε, αλλιώ πάλι δεν θα κάνουμε τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε πέντε εισαγγελείς και ε, ελεγκτές των λογαριασμών που εργάζονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιμένουν γιατί δεν αποζημιώνονται ούτε για τις δαπάνες τους και πραγματικά ε, πρέπει ε, να κάνουν ε, τρομερές οικονομίες. Είναι, είναι αναξιοπρεπές αυτό από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης θα πρέπει να δούμε πώς θα ενταχθούν στην ΕΙΕΔ ειδικοί εκπρόσωποι. αυτή είναι μια παλιά ιστορία επίσης που πάλι προσκρούει σε διάφορα ανόητα εμπόδια θα πρέπει να το τονίσουμε. Αυτό το έχει ζητήσει και το ελεκτικό συνέδριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενσωματωθούν οι ειδικοί αντιπρόσωποι εντεταλμένοι στην εξωτερική πολιτική. Δεν είναι πάρα πολύ πια, αλλά αυτοί που έχουμε θα πρέπει να ενταχθούν στην ΑΕΔ. Αλλιώ, έχουμε ε, τους πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικού απεσταλμένους, ε, ε, δεν μιλάμε με μία φωνή ε, στην εξωτερική μας παρουσία. Θα πρέπει όλοι αυτοί να ενταχθούν στην ΕΕΔ για να είναι κάπου ενταγμένοι. Το ξέρω ότι θα τσακωθείτε με το Συμβούλιο, αλλά αξίζει τον κόπο αυτός ο καυγάς για να έχει μια συντεταγμένη και ενωμένη παρουσία η Ένωση προς τα έξω. Αυτό ήταν το δεύτερο. Τρίτον, η Γενική Διεύθυνση για τα περιφερειακά κονδύλια διαχειρίζεται δισεκατομμύρια και σε δύσκολες χώρες ε, για τα ταμεία συνοχής. Έχουμε 50 οικονομικούς ελεγκτές που ασχολούνται σε αυτή τη Γενική Διεύθυνση με τον έλεγχο των συγκεκριμένων κονδυλίων. Μήπως θα μπορούσαμε να αυξήσουμε τις θέσεις για να κάνουμε κάτι να ελέγχουμε τα κονδύλια αυτά. Γιατί τελικά πραγματικά θα αξίζει τον κόπο κάτι τέτοιο. Αυτό δεν θα αρέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε κανέναν, αλλά τι να κάνουμε. Πιστέψτε μας ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό και για τις ίδιες χώρες. Δεν είναι δαπάνη, αυτό οικονομία είναι. Γιατί αν βοηθήσουμε από την αρχή τις χώρες δεν χρειάζεται να ανακτήσουμε τα χρήματα στο τέλος και να τους τα ξαναζητάμε. Δεν μπορούν να τα κρατήσουν δηλαδή. Αυτά από πλευρά μου. Δεν ξέρω συνάδελφοι αν θέλουν το λόγο. Ο Τάμας Σιτχόφσκι. Ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βιώτη που είναι σήμερα εδώ μαζί μας Νομίζω ότι είναι καλή ευκαιρία να έχουμε την ανταλλαγή απόψεων αυτή και η Ίγκε Γκρέσλε σας εξέφρασε την άποψη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εγώ θα σας παρουσιάσω μια άλλη οπτική γωνία. Την οπτική γωνία ενός ανθρώπου που ασχολείται με τον προϋπολογισμό για θέματα ασφάλειας στην ασφάλεια δεν έχουμε χρήματα για επιχειρήσεις ή για το Eurojust ή για εξοπλισμό. Το Eurojust ε, έχει ξεμείνει σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις του. Δεν μπορεί να φέρει σε πέρας ε, ε, τα καθήκοντά του, ούτε οι εισαγγελείς δεν μπορούν να συναντηθούν ελήψη χρημάτων. Και χρειάζεται παρόλα αυτά να αγωνιστεί κάποιος και κατά μέτωπον να αντιμετωπίσει το πρόβλημα γιατί είναι και ενοχλητικό και αναξοπρεπές. Ένας εισηγητής γνωμοδότησης αν πρότεινε αύξηση στον προπολογισμό και η αύξηση αυτή συναντούσε το βέτο της Επιτροπής Προπολογισμών δεν θα ήταν κάτι που θα χαροποιούσε αυτό τον εισηγητή φαντάζομαι. Εγώ και άλλοι που εργαζόμαστε στα θέματα αυτά είμαστε προσιλωμένοι στο έργο μας. Τέσσερα χρόνια τώρα δουλεύουμε πάνω σε αυτό το θέμα και γνωρίζουμε ποιοι εκτελεστικοί οργανισμοί κάνουν καλή δουλειά και ποιοι όχι και νομίζω ότι οι προτάσεις μας ε, είναι σωστές. Έχω διαβάσει τις παρατηρήσεις ε, και την παρουσίαση που θα υποβάλλετε. Δεν ξέρω αν έχετε δει την απαλλαγή του 2016 για την Κομισιόν και τους ε, εκτελεστικούς οργανισμούς. Εκεί επισημάναμε πάμπολα προβλήματα, περιπτώσεις ε, κακής ε, ε, διαχείρισης και διασπάθησης κονδύλιων. Είχαμε σήμερα στην Μέσια διάταξη και δύο ειδικέ εκθέσεις που δείχνουν ότι δεν μετράτε παρκώς το αποτέλεσμα των δαπανών αυτών. Έχουμε ποσοτικούς στόχους και μετράμε το πόσα πράγματα έχουμε χωρίς να, χωρίς να υπολογίζουμε την ποιότητα και την προσθέμενη αξία στις εκάστοτε περιοχές. Να σας δώσω ένα παράδειγμα από την περιφερειακή ανάπτυξη. Προτείναμε 100 εκατομμύρια για την Τσεχία. για να φτιάχνουν τα τοπίο ε, τα τοπία καλύτερο ψωμί, τα τοπία που προμηθεύουν ε, τον Πρωθυπουργό. Μα είναι γελίο κάτι τέτοιο. Συγκεκριμένα να υποστηρίξουμε ένα αρτοπίο, ενώ υπάρχει δίπλα ένα άλλο που μπορεί να κάνει το ίδιο και πιο αποτελεσματικά, χωρίς να επιδοτείται από την Ένωση όμως. Τέτοια πράγματα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Είναι πολύ σημαντικό όταν θα έχετε επαφέ με τα κρατημέλη να τονίζετε ότι αυτό που απαιτείται είναι τα αποτελέσματα, η αποτελεσματικότητα. Και η αύξηση των ελεγκτών είναι κάτι πολύ αναγκαίο. Για την περίπτωση της Τσεχίας έχουμε την υπόθεση του λεγόμενου Storknest, μιας επιχείρησης. Δεν ανακαλύφθηκαν τα προβλήματα και τα σκάνδαλα παρά από την όλα. Τόσο χρειάστηκε να περιμένουμε. Ο κύριος Βον. Καλωσορίζω τον κύριο Βιώτη. Έχει σημαντική ε, δουλειά να κάνει στο Κοινοβούλιο και νομίζω ότι τα καταφέρνει καλά μέχρι στιγμής. Και οι προτεραιότητες που έθεσε για τον προϋπολογισμό, βιωσιμή ανάπτυξη, καινοτομία, κλιματική αλλαγή, μετανάστευση, ασφαλή κτλ. μας βρίσκουν σύμφωνος. Είναι καλές προτεραιότητες. Επίσης η προτεραιότητα που ανέφερε για την ανεργία των νέων και αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό. Και γνωρίζουμε στην Επιτροπή μας ε, και το Λεκτικό Συνέδριο αλλά και εμείς ε, έχουμε ερευνήσει την εγγύηση για την νεολαία για παράδειγμα και ε, καλό είναι να δούμε τι μπορεί να γίνει, γιατί ξεκινήσαμε πολύ αργά και πρέπει να ε, επιταχύνουμε για το μέλλον. Αν εσεί δεν μπορείτε να μελετήσετε τα συγκεκριμένα θέματα, ίσω μπορούν ε, οι συνεργάτε σα. Μίλησαν συνάδελφοι για τι ειδικέ εκθέσει. 3,1% έχουν μειωθεί τα ποσοστά ασφάλματο στην τελευταία αίτησια έκθεση. Το διαβάζουμε αυτό. Υπάρχουν όμω κάποιε ανησυχίε η πολιτική συνοχή σε μένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ ε, και η περιφερειακή ανάπτυξη είναι θέμα. Θα πάτε σε αυτή την επιτροπή αύριο. Έχουμε χαμηλά ποσοστά εφαρμογής σε ορισμένα κράτη-μέλη. Άρα ό,τι κάνετε εσείς ε, είναι ουσιαστικά ε, η κατάρτιση του προπολογισμού του τελευταίου έτου του τρέχοντος απολύτως μεσονομικού πλαισίου. Πρέπει να δαπανηθούν τα κονδύλια της συνοχής τώρα και για τα σωστά, γιατί αλλιώς θα δοθεί πρόσχημα και δικαιολογία σε όσους θέλουν να κόψουν τα κονδύλια συνοχής να, τα, να το κάνουν στο προσεχές πολιετές ονομικό πλαίσιο. Ξέρω ότι όσοι εισηγητή για τον προβλησμό δεν είναι εύκολα πιέσετε τα κρατημέλη να κάνουν δαπάνες, Αλλά ασκήστε όλοι σας την επιρροή παρακαλώ, ώστε τα κονδύλια της συνοχής να δαπανηθούν μέχρι το τέλος ε, ισχύω του τρέχοντος ε, πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου για να μην έχουν δικαιολογίε για να περικόψουν τα κονδύλια όσοι το θέλουν αυτό. Ο κύριος Τσέλερ, ο οποίο έχει αναλάβει τη στέξη νομοδότησης ε, για εμά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Δεν άκουσα τον κύριο Βιώτη, αλλά ήμουν στην Περιφερειακή Επιτροπή και ο συνάδελφο Βόν αναφέρθηκε μόλι αυτό. Εκεί ε, κατά κύριο λόγο το θέμα είναι πώς θα σώσουμε τα κονδύλια για τη διορθωτική πολιτική και το Ταμείο Συνοχής και πώς θα ε, συνδυαστούν τα εργαλεία αυτά και τα μέσα για να μπορούν να αποδίδουν και μετά το 2020. Και τι θα γίνει με τα ποσά που είναι στους εθνικούς φακέλους και πώς μπορούμε να τα συνεχίσουμε, να τα χρησιμοποιούμε στο μέλλον αλλάζουν και κάποιες νομικές βάσεις και κάποια νομοθεσία. και αυτό θα έχει επιπτώσεις στον προπολογισμό του 2019, που είναι το πρώτο τελευταίο έτος της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να συζητήσουμε ε, τα όσα έχουμε επικρίνει ε, σε προηγούμενες εκθέσεις απαλλαγής, ε, στρεβλά στη Γεωργία, το πρόγραμμα για το πρασίνισμα ή το πρόγραμμα για τους νέους αγρότες, τι θα τα κάνουμε αυτά. Είτε θα τα βοηθήσουμε να αποδώσουν, είτε αν αποδειχθούν ατελέσφορα και δύσκολα στην εφαρμογή τους, να δούμε τι θα κάνουμε και πώς θα διοχετεύσουμε τα κονδύλια σε άλλους διάβλους εκεί που αποδίδουν και πιάνουν τόπο. Στην αναπτυξιακή πολιτική τώρα έχουμε κάποια καταπιστεύματα που θα αρχίσουν να δουλεύουν, όπως μας διαβεβαίωσαν οι συνάδελφοι από την Επιτροπή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Αυτά τα καταπιστευματικά ταμεία, έτσι ώστε θα να απορροφήσουν πόρους. Αυτό τον καιρό έχουμε τη διάσκεψη των δωρητών για τη Συρία, όπου τάζουν δισεκατομμύρια για την ε, ανοικοδόμηση, μάλλον την ε, ανασκρότηση τη χώρας για να επιστρέψουν και οι πρόσφυγες. Πού θα τα βρουν τα λεφτά, από τα κράτη-μέλη ή μήπω από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπω έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν σε διάφορα κονδύλια. Και πόθεν από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Γιατί υπάρχει το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο που δεν προβλέπει τέτοια κονδύλια τα πήραν από αλλού, από άλλες γραμμές του προπολογισμού. Και μάλιστα ξύνοντας διάφορα σερτάρια και υπολείμματα για να τα συγκεντρώσουν. Ναι, αλλά αυτά τα χάνουν οι αρχικές πολιτικές. Είτε πρόκειται για τη Γεωργία, την Αλία ή την πολιτική συνοχής. Που συνήθως είναι τα πρώτα θύματα. Το είπε και ο Ντέρεκ Βον Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη όπου η φάση της εφαρμογής δεν είναι ακόμα ικανοποιητική. Μετά από 5-6 χρόνια της υλοποίησης και της εκτέλεσης των διευθυντικών ταμείων. Συναρπαστικό το εγχείρημα. Και έρχεται και η συζήτηση για το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο να αντιταχθεί σε αυτό που για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και το τρέχον πλαίσιο δεν έχουμε καν μια λογική ενδιάμεση μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση. Καλή επιτυχία κύριε Βιώτη. Είδαμε ποιες είναι οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές και τα κέντρα βάρους για τον προϋπολογισμό του 2019 και από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού σίγουρα θα κάνουμε και κολλιά μας και τη γνωμοδότησή μας. Ο κύριος Ωρέλα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Uh, Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ ε, σημαντική αυτή η ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Βιώτη, τον εισηγητή. εμεί. Ε, Ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώσαμε προσεκτικά και τι παρατηρήσει τι δικές του, αλλά βεβαίω και τι παρατηρήσει που έκαναν τα μέλη τη Επιτροπή, και φυσικά θα μεταφέρομαι ακριβώ αυτή την ανταλλαγή θέσεων στην Επιτροπή όσον αφορά την τελευταία, ε, το τελευταίο σχόλιο παρατήρηση του κυρίου ε, Τσέλερ και εγώ ρώτησα, υπέβαλα την ίδια ε, ερώτηση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών χθες. Από όσο καταλαβαίνω, στη διαδικασία αυτή, τη διαδικασία που, έχει, που τώρα λαμβάνει η χώρα, η Κομισιόν έχει υποβάλει ε, ένα αίτημα ε, αντίστοιχο αυτού που είχε κάνει τον προηγούμενο χρόνο. Είχε κάνει μία έκκληση ε, για... Last 560 εκατομμύρια ε, και νομίζω ότι το ίδιο ζητάμε και για τον, ε, το 2019 ε, έτσι όπως θα εμφανιστεί στον, στον που θα εκδοθεί τον Μάιο και θα δημοσιευτεί. Πρόκειται να υπάρξει μία, ένα μείγμα από καινούρια χρήματα αλλά και από αναμόχληση παλαιών αχρησιμοποιητών κονδυλίων. Όσον αφορά δε την κατανομή θα αποφασιστεί αργότερα. Ευχαριστώ κύριος Βιώτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, που ε, προκάλεσαν μια πάρα πολύ χρήσιμη ε, συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Εγώ σημείωσα όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν και για τη Eurojust και για την Όλαφ, καθώς επίσης και τους προβληματισμούς για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, για τη Συρία, για όλα. Τα έχω λάβει υπόψη μου, όπως έκανα άλλωστε και με τις άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ευχαριστώ τον Σάιφο Βόγαν. Ε, διότι αναφέρθηκε στην έκθεση για την ε, εγγύηση των νέων, Youth Guarantee, καθώς επίσης και για την ανεργία των νέων. Ε, οι συνάδελφοι επίσης συζήτησε το θέμα μάλλον και με τις συναδέλφους της Επιτροπής ΕΜΠΛ γιατί πραγματικά εγώ γνωρίζω την εργασία σας και την εκτιμώ ιδιαίτερος. Αυτή τη στιγμή δεν έχω ιδιαίτερες παρατηρήσεις να κάνω, γιατί η έκθεσή σας, ε, η επιστολή σας ε, θα προκύψουν και θα τις λάβω υπόψη μου. Αυτό που επαναλαμβάνω είναι ότι πρέπει να εργαστούμε από κοινού και αν μπορώ να δώσω μια συμβουλή ε, σαν φίλος και όχι σαν εισηγητής για τον προπολογισμό. συχνά τα προβλήματα, για να μην πω πάντα, τα προβλήματα προκύπτουν στο Συμβούλιο. Εάν κάποιος από εσά μπορεί να ξεκινήσει να δουλεύει το θέμα και να προετοιμάζει τις χώρες σας πριν από τη διαβούλευση... Ε... πριν από τη συνδιαλλαγή, συγγνώμη, ε, καλό θα ήταν. Ε, αυτό είναι η πιο καυτή πατάτα τώρα, πώς να το πω. Θα κάνουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε. Ξέρω ότι κι εσείς κάνετε ό,τι μπορείτε, δεν είναι και εύκολη δουλειά σας. Ε, θα σας στείλουμε τη γνωμοδότηση και θα παλέψουμε μέχρι τελευταία στιγμή. Είναι ένα θέμα πολύ κουραστικό ε, και ε, είναι πολύ καλό να έχουμε ένα εισηγητή που παλεύει και αυτό. Σας ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Επομένως, ολοκληρώθηκε αυτό το σημείο της διάταξης και περνάμε στο 12 την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Παρθμών 9 του 2018. Ο Λιμπεράτσκι είναι ο και έχουμε και τον κύριο Χέριξ από το, αρμοδιο... από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι βουλευτές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση ε, να σας παρουσιάσω την έκθεση ε, του Ελεκτικού Συνεδρίου για τις, ε, δημόσιες, τις συμπράξεις τομέα να σας πω πρώτα απ' όλα ε, κάποια εισαγωγικά. Από το 1990 περίπου 1750 σχέδια συμπράξεων ε, δημοσιοδικού τομέα είχαμε αξία συνολικής 336 δισεκατομμυρίων ευρώ και στις περισσότερες περιπτώσεις στον τομέα των μεταφορών το 2016 αυτό ήταν το 1 τρίτο των ε, προγραμμάτων. Η οικονομική τώρα σημασία μειώνεται από το 2000 έως το 2014 μόνο 84 τέτοια σχέδια και πήραν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 5,6 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το 2015 Πλέον υπάρχει δυνατότητα για αυτά τα σχέδια να χρηματοδοτούνται και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το ΕΦΣΙ ή ΕΤΣΕ στα ελληνικά. Θα ήθελα τώρα να έρθω σε κάποιες συστάσεις, αλλά ε, πρώτα να μιλήσω και για ε, το σχεδιασμό ε, και στα θεσμικά ζητήματα να αναφερθώ. Υπάρχουν πραγματικά κάποιες ελλείψεις και στο νομικό και στο θεσμικό πλαίσιο και τις σχετικές διαδικασίες. Για παράδειγμα, δεν υπάρχουν σαφείς πολιτικές έννοιες, ιδέες και στρατηγικές για τη χρήση ε, των συμπράξεων αυτών. Τι κάνουν δηλαδή αυτά τα προγράμματα, πώς χρησιμοποιούνται τα σχετικά κονδύλια. Ε, το ελεκτικό συνέδριο στις περισσότερες ε, χώρες δεν έχει συγκεντρώσει, βλέπω ότι δεν υπάρχει επαρκής εμπειρία και δεν υπάρχει επίση επαρκής διοικητική ικανότητα των αρμόδιων αρχών σε ό,τι αφορά την υλοποίηση σχεδίων στον δημοσιοδικού τομέα. Υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο κίνδυνο ε, να υπάρξει μια αντιπαράθεση, μια αντίθεση και σύγκρουση αυτών των σχεδίων με την έμφαση που δεν όλο και περισσότερο η Ένωση ε, στο λεγόμενο, στη λεγόμενη μόχλευση. Ε, δηλαδή δεν κινητοποιούνται τελικά επαρκή ιδιωτικά κεφάλαια. Ποιες είναι τώρα οι συστάσεις μας ε, για την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη καταρχάς. Ε, δεν ε, θα πρέπει να προχωρήσουν σε πιο εντατική ε, ενίσχυση αυτών των προγραμμάτων όσο παραμένουν τα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει. Η Κομισιόν τώρα θα πρέπει να παρέχει χρηματοοικονομική υποστήριξη σε αυτές τις ε, κοινοπραξίες μόνο όταν έχουν υψηλή στρατηγική σημασία και συνάδουν με, με σαφείς πολιτικές δεσμεύσεις και στρατηγικές για τους τομείς που είναι οι πλέον κατάλληλοι για την ε, αξιοποίηση αυτών των ε, σχεδίων. Σε ό,τι τώρα την αξιολόγηση αυτών των σχεδίων, Έχουμε περιγράψει και προειδοποίησει για τον κίνδυνο που μπορεί να υπάρχει. Ε, Παραδείγματο χάρη, ε, ο περιορισμός της δράσης των ε, αναθετουσών αρχών ε, και κάποια δυσανάλογα αποτελέσματα. Πολλές φορές υπογράφονται συμβάσεις προτού ξεκαθαρίσουν ε, σημαντικά ζητήματα. Παραδείγματο παραδείγματος χάρη, τι γίνεται με τη χρήση γης, τι γίνεται με δυνατές ενδεχόμενες απαλυτρώσεις κτλ. Επίσης είδαμε να υπάρχουν καθυστερήσεις ό,τι αφορά την εφαρμογή 7 από τα 9 ε, σχέδια σε Γαλλία, Ελλάδα, ε, Γαλλία, Ελλάδα και Ισπανία 5-20 μήνες. Επίσης σημαντική αύξηση του κόστους παρατηρήσαμε, δηλαδή χρειάστηκαν 1,5 δισεκατομμύρια πλέον δημόσια κονδύλια για την ε, ολοκλήρωση αυτών των προγραμμάτων, 1,2 δίσε στην Ελλάδα και 0,3 δις στην Ισπανία και το 30% των ποσών αυτών ε, είχαν διατηθεί από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Άρα δεν είχαμε αποτελεσματικές δαπάνες και αυτό ε, αποτελεί δεδομένο για το 20%. Ε, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ανέφερα την Ελλάδα γιατί το 59% ε, ε, το 3,3 δις ευρώ πηγαίνουν στις στη χώρα αυτή, 5,6% μόνο σε Γαλλία και Ισπανία. και ε, για τους αυτοκινητόδρομους έχει αυξηθεί σημαντικά το κόστος από ε, το 59% στο 69%. Και το κόστος ε, αναχιλιόμετρο είναι ένας δείκτης πάρα πολύ σημαντικός 69% όπως είπα ήταν η αύξηση και αυτό είναι πολύ σημαντική επιβάρυνση για την κατασκευή του οδικού δικτύου. Και τα κράτη-μέλη λοιπόν θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ε, τις ε, ε, νέες διαπραγματεύσεις και τις καθυστερήσεις, πόσο κόστος επιπλέον μπορεί αυτό να συνιστά. Θα πρέπει λοιπόν να μειωθεί το επιπλέον κόστος και θα πρέπει οι διαπραγματεύσεις να γίνονται έγκαιρα και αναδιαπραγματεύσεις των σχετικών συμβάσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επιλογή. Ε, πολλές φορές γίνεται χωρίς να έχουν γίνει συγκρίσεις και αναλύσεις αναλλακτικών λύσεων. Αυτό το είδαμε στην Ισπανία και στην Ελλάδα. Ε, ενώ Γαλλία, Ιρλανδία, εκεί ε, διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε ανάγκη, τέλο πάντων δεν υπήρχε κάποια διάταξη που να επέβαλε την ανάλυση αυτή. Και σε ό,τι αφορά την επιλογή που επελέγει. Δεν ξέραμε κατά πόσο ήταν η καλύτερη επιλογή σε ό,τι αφορά ε, το κόστος ε, ε, και την αποτελεσματικότητα. Επίσης, πολλές φορές ήταν πάρα πολύ αισιόδοξα τα σενάρια τα οποία επελέγησαν, η επιλογή δηλαδή που Και παραδείγματος χάρη στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών ήταν κάτω από τις προγνώσεις Ιρλανδία, δηλαδή, Γαλλία, κατά 69, 69 κατά 69%. Ε, στην Ελλάδα ε, επίσης αρνητικά ποσοστά είχαμε και σε άλλες χώρες. Επίσης, ό,τι αφορά την ανάλυση κινδύνου, πάλι εδώ δεν είχαμε ε, συνεκτικές και αποτελεσματικές διαδικασίες με αποτέλεσμα να έχουμε ή υπερβολική εκτίμηση ή πολύ χαμηλή εκτίμηση των κινδύνων. Δεν ελήφθησε λοιπόν, δεν ελήφθη αυτό σωστά υπόψη το γεγονός. Κάτι άλλο το οποίο είδαμε. Ε, είδαμε τον κίνδυνο να υπάρχουν κάποιες αρνητικές ε, παρενέργειες ε, εκτός των ισολογισμών είχαν καταγραφεί αυτά τα σχέδια και η αρχή της διαφάνειας δεν ελήφθη επαρκώς υπόψη. Και δεν ελήφθησαν επικώ υπόψη επίση ε, τα χρέη και υποχρέωση των κατομελών τι επιπτώσει θα είχαν. Ζητούμε λοιπόν σε σχέση με αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέχει υποστήριξη σε τέτοια σχέδια μόνο αν είναι βέβαιο ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι δημοσιονομικές παράμετροι ε, και οι οικονομικές παράμετροι για την επιλογή αυτών των σχεδίων και να μην υπάρχουν ε, κάποια άλλα στοιχεία, στατιστική επεξεργασία ή προσωπική περιορισμοί που να επηρεάζουν και βέβαια θα πρέπει ε, να έχουν προηγηθεί στέρες και συγκριτικές αναλύσεις. κατακλείδη διαπιστώνουμε ότι αυτές οι συμπράξεις ε, δημόσιο-δυτικού τομέα, τα ΣΔΙΤ αυτά, ε, παρουσιάζουν ελλείψεις και ε, γι' αυτό θεωρούμε ότι δεν φέρνουν επαρκή ωφέλη, αλλά αντίθετα παρουσιάζουν πολλά μενικτήματα. Πρόεδρος, εισηγητής ο κύριος Λιμπεράς, παρακαλώ. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. If you're permission, may I speak Polish? Ευχαριστώ. Μπορώ να μιλήσω στα, στα πολωνικά. Ήταν πάρα πολύ ε, ευχάριστο που συνάντησα την ομάδα από το ελεγκτικό ε, ε, συνέδριο. Πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και πρέπει να πω ότι πρόκειται εδώ για ένα εξαιρετικό έγγραφο βασίζεται δε ε, σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε πολύ συγκεκριμένα ε, στοιχεία ε, και μπορώ ως γενική γραμμές να συμφωνήσω με τις συστάσεις. Έχω και κάποιες επιπλέον συστάσεις, εγώ ο ίδιος. Στη δική μας Επιτροπή, αλλά και στην Επιτροπή Μεταφορών, πριν από λίγα χρόνια, αναρωτιόμαστε εάν και εφόσον θα έπρεπε να υπάρξουν συγκεκριμένες κατευθυντήρες γραμμές ή ίσως και κάποια οδηγία ε, σχετικά με το πώς ε, να γίνονται αυτές ε, οι συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, η PPP. Και είχαμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το ενδιαφέρον του δημοσίου ε, μάλλον το συμφέρον του δημοσίου ε, τομέα θα έπρεπε να ληφθεί περισσότερο υπόψη. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ε, κάποια επίκριση τις ε, τάσεις ε, που έχει ο δημόσιος τομέας ε, να περιφρονεί το δημόσιο καλό και να χρηματοδοτεί κάποια πολύ περίεργα και εξεζητημένα προγράμματα τα οποία θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις εκλογές ή δεν ε, παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Διαπιστώνουμε ότι και η διαχείριση κινδύνου είναι ασθενής ε, και ο πολιτικός κίνδυνος επίσης δεν λαμβάνεται σωστά υπόψη. Αυτό το διαπιστώσαμε στην Ελλάδα, όπου μια νέα κυβέρνηση οπισθοχωρεί όσον αφορά τις δεσμεύσεις της προηγούμενης κυβέρνησης και δεν είναι μάλιστα και η μόνη κυβέρνηση. Ε, πρέπει να γίνονται σωστές αναλύσεις κόστους αποτελεσματικότητας. Ε, και για τον ε, δημόσιο εταίρο και για τον εταίρο που προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα και οπωσδήποτε ε, monitoring σε πραγματικό χρόνο ε, και δυνατότητα αντίδρασης σε κάθε περίπτωση. Δεύτερον, το χρονοδιάγραμμα ε, συχνά δεν ε, οργανώνεται σωστά όσον αφορά την επιστροφή, την απόδοση ε, της επένδυσης και συμφωνώ με το σχόλιο που ακούστηκε ότι πολλές φορές τα προγράμματα γίνονται με καλό σκοπό και καλή πρόθεση αλλά αντί να γίνουν ακριβώς τα πράγματα όπως έπρεπε να γίνουν έτσι ώστε να έχουν καλή, καλή απόδοση αποφασίζεται ενδιάμεσα να γίνει κάτι πολύ πιο μεγάλο και πολύ πιο δαπανηρό και εν τέλει η ε, επιστροφή δεν επιτυγχάνεται. Όσον αφορά την Κομισιόν, πολύ συχνά ακούμε από πλευράς της Κομισιόν «αυτό δεν αφορά την Κομισιόν». Αυτό είναι θέμα αποκλειστικής αρμοδιότητας των κρατών μελών, δεν μπορεί να αναμειχθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και φτάνουμε σε σημείο να αναρωτιόμαστε, «Ε, και στο τέλος τι κάνει η Κομισιόν, τι χρειαζόμαστε μια τέτοια Κομισιόν, εάν δεν μπορεί να αναμειχθεί η Κομισιόν, εάν είναι απ' έξω και παρακολουθεί μονάχα τα πράγματα ως παρατηρητής, τότε θα πρέπει, χρειάζεται ε, ε, αλλαγή των συνθήκων 500 δις ευρώ ε, ε, για το ΕΦΣΥ. Και ένα μεγάλο κομμάτι ε, θα πάει σε μεγάλα προγράμματα. Απ' την άλλη μεριά έχουμε και τους ιδιωτικούς επενδυτές, αυτούς που είναι από την Κεντρική Τράπεζα, αυτούς που προτείνει η Τράπεζα Επενδύσεων και ένα σωρό άλλα πράγματα. οπωσδήποτε θα πρέπει όλες οι πολιτικές να είναι συνεκτικές μεταξύ τους. Ε, γιατί αυτό που θέλουμε είναι μια πραγματική συνοχή στην Ευρώπη και μια πραγματική ε, βιομηχανική επανεκκίνηση της Ευρώπης. Ε, η έκθεση αυτή είναι ορθή, έρχεται την κατάλληλη στιγμή και τα ευρήματα τα οποία προκύπτουν από αυτήν είναι πολύ σημαντικά και θα πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε τρόπους για να λυθούν τα προβλήματα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί στην έκθεση αυτή. Και θα ήθελα η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σταματήσει να χώνει το κεφάλι της στην άμμο και να δει τα πράγματα κατά πρόσωπο. Ευχαριστώ. Ε, σύντομη παρουσίαση είπαμε. Αλλά βεβαίω θέλουμε να δώσουμε και το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τη Γενική Γραμματεία, να μας πείτε και το δικό σας ρόλο στι αποφάσεις αυτές για τις ΣΔΙΤ. Και δεν σας βλέπω. Πού είστε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ που μας καλέσατε στη σημερινή συζήτηση για ένα τόσο σημαντικό θέμα που αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο δημόσιο τομέα μπορεί να υποστηρίξει τι επενδύσει με διάφορου τρόπου. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να πω ότι συμμεριζόμαστε μερικά από τα συμπεράσματα ε, της έκθεσης. Βεβαίως, η εμπειρία από τη ΣΔΙΤ είναι μεικτή, ένα μεικτή στην Ευρώπη, εξαρτάται πάρα πολύ από το κράτος μέλος και από τον εκάστοτε κλάδο. Ε, είναι σημαντικό ιδιαίτερα να εστιάσουμε πάρα πολύ ε, στις τεχνικές δυνατότητες. Δηλαδή, ε, για να προχωρήσει ένα έργο από τη σύλληψή του μέχρι την εκτέλεσή του, εξασφαλίζοντας ότι θα πιάσουν τόπο τα χρήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι ιδιαίτερα προσιλωμένη στι ΔΙΤ. Αυτό είναι ένα μοντέλο μεταξύ άλλων. Οι συμπράξει δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Είπαμε ότι είναι ανάμεικτη εμπειρία. Πάντω έχει λειτουργήσει καλά σε πολλά κράτη-μέλη. Και σε ορισμένα κράτη-μέλη επίση επέτρεψε να γίνουν έργα ε, επωφελή και να έχει κέρδος και το δημόσιο. Αναφέρθηκε το σχέδιο επενδύσεων για την Ευρώπη και ακριβώς εκεί υπήρχε ένας πυλώνας ξεχωριστός για την τεχνική βοήθεια και υποστήριξη ε, στις δημόσιες αρχές. Αυτό έχει εφαρμοστεί ε, στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και είχαμε αρκετά καλά παραδείγματα. Άλλο σημαντικό στοιχείο που αξίζει να αναφερθεί είναι το εξής. Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη δεν αφορά μόνο μεγάλα έργα υποδομών, έχει δύο θηρίδες επενδύσεων. Και η μισή στήριξη πηγαίνει σε εταιρείε μικρομεσαίες και μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Καταλήξαμε ότι οι ΣΔΙΤ επέτρεψαν να γίνουν μεγάλα έργα υποδομών και τις περισσότερες φορές είναι καλή επιτήρηση και η συντήρηση. Σε ό,τι αφορά τις προθεσμίες και τις καθυστερήσεις, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι υπήρξε η κρίση δημοσίου χρέους και η ύφεση που επηρέασε ε, πολλά από τα κράτη-μέλη όπου έγιναν οι έλεγχοι και αυτό μπορεί να εξηγήσει εν μέρη την καθυστέρηση που σημειώθηκε. Ποιος ευθύνεται τώρα μάλλον ποιος φέρει την ευθύνη να αποδώσει εις ΔΙΤ, το κράτος μέλος. Ε, θέλω και πάλι να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι πολύ ε, ε, καλή αυτή η προσπάθεια και αυτή η εμπειρία και πραγματικά ορισμένε ΔΙΤ πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Ναι. Τώρα θα καταλάβετε ότι δεν μας ικανοποιούν αυτά που μας είπατε. Πέρα από το γεγονός ότι είναι μία από τις περιπτώσεις αυτές όπου ε, ε, είναι μια αδικία. Έχουμε εδώ τμήματάρχη που ε, ακούει τα σχολιανά του. Το έχουμε γράψει στην ημερήσια διάταξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εδέησε να έρθει στο αντίστοιχο επίπεδο υπαλλήλου εδώ. Εγώ δεν θέλω να σας κατηγορήσω για τίποτα, αλλά είναι άδικο που σας έχουν στείλει εσάς εδώ. Εντάξει, αν δούμε την έκθεση, πήγαν στραβά κάποια πράγματα. Μόνο ε, στραβά, έχουμε δραματικές εξελίξεις και ανευθυνότητα. Ανευθυνότητα, τι έγινε, τρέχουν από τα πατζάκια μας τα λεφτά και δεν τα προσέχουμε στον τρόπο με τον οποίο τα δαπανούμε. Και αυτό το έχουμε δει από παλιά. Στη δική μου περιφέρεια πριν από 20 και 25 χρόνια φτιάξανε μια σύραγγα ε, στο Engelberg με ΣΔΙΤ. Τα, ξέρει ο Επίτροπος τότε γιατί κυβερνούσε. Αποτέλεσμα. 25% ακριβότερη ΣΔΙΤ από αν ήταν δημόσια η επένδυση. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε τέτοια στρεβλή εξέλιξη για τέτοια τρομερά ποσά. Θα θέλαμε αυτές τις ερωτήσεις να μας τις απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτενώς και να ακούσουν και το τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολείται ε, με τα διδάγματα του παρελθόντος. Και το να μου λέτε ότι δεν φταίμε εμείς και δεν ήταν δική μας ευθύνη, τι να πω, δεν με ικανοποιεί καθόλου. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά τόσο σημαντικά πράγματα με τέτοια επιπολαιότητα και να τα διεκπεραιώνουμε. Εντάξει, δεν πήγανε καλά και τι να κάνουμε. Όχι, θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ για τα όσα είπατε. Ε, ζητώ συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να μας ξανάρθετε. Έχουμε και δεύτερο γύρο. Τώρα αυτή ήταν μια σύντομη παρουσίαση. Πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Επίζω και οι αρμόδιες ε, επιμέρους επιτροπές να επιληφθούν. Τουλάχιστον η Επιτροπή Μεταφορών παρακαλώ να προσέξει τη συγκεκριμένη έκθεση και να το συζητήσει. Έχετε, κύριε Γέριξ, ε, ε, προσκλήσεις από τις άλλες επιτροπές. Όχι. Η Επιτροπή Μεταφορών σήμερα έχει προσκληθεί, αλλά τι να κάνουμε να του στείλουμε την έκθεση για να τη διεκπαιρεώσουν και αυτοί. Ευχαριστώ και πάμε στο επόμενο θέμα. Ε, κύριε Χέριξ, ε, ε, Α, και η Επιτροπή Προεπολογισμών λέει ο κύριο Τσέλερ. Βεβαίω, και η Επιτροπή Προεπολογισμών. Ευχαριστώ. Uh, thank you. Let's go on to item uh, 13, which is the να πάμε στο 13 ειδική έκθεση για την ανανεώσιμη πηγές ενέργεια λοιπόν για βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη τι δυνατότητες ενεργειών παραμένουν πολύ σαν χρησιμοποιητέ. Ε, κύριε Κάντε, Μάρχη, είναι εισηγήτρια, αλλά έχουμε τον κύριο Γέρεμπε εδώ, τον θα πάρει καταρχά το λόγο. Ευχαριστώ αγαπητοί ε, ευρωβουλευτές μου δίνετε το λόγο για να συζητήσουμε τα βασικά απορίσματα τη ειδική μας έκθεσης στην χρήση ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη. Πολλοί ε, πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δοθεί έτσι ώστε να προωθηθεί η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεταξύ των οποίων ε, και το ε, Ταμείο για τη Γεωργική Ανάπτυξη. Εμείς μελετήσαμε το πλαίσιο πολιτικής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σύνολο της πολιτικής για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, είδαμε και μελετήσαμε πώς την επίδοση που έχουν τα προγράμματα με ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και είδαμε ότι μπορεί να υπάρχουν συνέργειες ανάμεσα στις ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας και τα υπόλοιπα ε, προγράμματα που αφορούν την ανάπτυξη της ε, υπαίθρου αλλά δεν χρησιμοποιούνται όσο γίνεται, δεν χρησιμοποιούνται στην πλήρη τους δυνατότητα. Θα πρέπει οπωσδήποτε για να φτάσουν να αποδώσουν όπως πρέπει να βασίζονται σε συγκεκριμένη πολιτική βάση των ειδικών χαρακτηριστικών χαρακτηριστικών ε, των συγκεκριμένων ε, περιοχών. Ε, θα πρέπει επίσης να υπάρχει συνδυασμός και, το, και με τα εθνικά προγράμματα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης προέκυψε ότι ορισμένα εργαλεία στο πλαίσιο πολιτικής για τις ανανεώσιμες πηγές έχουν την δυνατότητα να βελτιώσουν την κατάσταση. Αλλά ούτε το ε, τωρινό ούτε το μελλοντικό πρόγραμμα στήριξης της, ε, των ε, άλλων μορφών ενέργειας δεν έχουν λάβει υπόψη όλους του, όλα τα στοιχεία, κοινωνικά, οικονομικά κλπ, έτσι ώστε να μπορέσουν πραγματικά να υποστηρίξουν την ανάπτυξη. τα, κύρια προβλήματα αφορούν την εντατικοποίηση της γεωργίας, καθώς επίσης και την καύση των βιο της βιομάζας ε, και ε, αυτό δημιουργεί ε, προβλήματα όσον αφορά την χρήση την, της εκπομπές καθώς επίσης και την αδυναμία αντιμετώπισης τους επίσης η σωστή ανάπτυξη της επέθρου θα πρέπει οπωσδήποτε να παίξει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για, την, για τις ανανεώσιμες ε, πηγές. Ωστόσο η Κομισιόνα δεν έχει δώσει αρκετές ε, διευκρινήσεις, διευκρινήσεις ούτε έχει πει με ποιο τρόπο ε, θα προκύψουν αυτές οι συνέργειες ή οι συνδυασμοί ανάμεσα στο πρόγραμμα για τις ανανεώσιμες και το πρόγραμμα για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Ενώ κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει αβιώσιμη μια ανάπτυξη στην ε, Ήπεθρο. Ωστόσο, έχουμε δει και κάποια καλά παραδείγματα καλής ε, πρακτική όπου έχει χρησιμοποιηθεί σωστά η κοινή στρατηγική. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2017, τέσσερα χρόνια δηλαδή σχεδόν, μετά από το ε, Μονάχα, ε, τέσσερα χρόνια δηλαδή μετά από την έναρξη του παρόντος δημοσιονομικού πλαισίου, μονάχα 40 από τα 800 εκατομμύρια έχουν χρησιμοποιηθεί ε, και ε, επομένως είναι πάρα πολύ μικρά τα αποτελέσματα, πενιχρά τα αποτελέσματα και επίσης και η επιτήρηση και η παρατήρηση παρακολούθηση των προγραμμάτων δεν είναι ικανοποιητική. Ε, όσον αφορά δε την προγραμματική περίοδο για την ανάπτυξη της υπαίθρου, ε, επίσης δεν έχει προκύψει συνδυασμός με το ε, MFF. Επίσης δεν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με το πώς ακριβώς έχουν δαπανηθεί τα κονδύλια. Το 2014 για την περίοδο μέχρι το 2020 εξακολουθεί να παραμένει η ελληπής επιτήρηση, κυρίως λόγω των πολύ ε, ε, των πολύ περιορισμένων δικτών ε, επίσης ε, υπάρχουν ε, προβλήματα όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά σε διάφορες περιοχές στόχους. Η παρακολούθηση των προγραμμάτων, των προγραμμάτων αυτών σε σχέση και με την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών δεν είναι η ιδέουσα. Θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα, συγγνώμη, εκθέσεις αξιολόγησης, αλλά δεν αποτελούν από μόνες τους αξιόπιστο ε, εργαλείο θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ε, η ε, δυνατότητα ε, να υπάρχει μια, μια ενιαία αντιμετώπιση για αυτούς που παράγουν ενέργεια για την δική τους κατανάλωση ή για να πουλήσουν την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης είδαμε ότι στην, σε, κοντά σε περιόδους εκλογών είχαμε ε, γενικώ μία αύξηση κάποιων προγραμμάτων τα οποία λίγο αντίκτυπο είχαν όσον αφορά τις ανανεώσιμε πηγές ενέργειας και ίσως λίγο περισσότερο όσον αφορά ε, την τοπική ε, οικονομία. Δεν παρατηρήσαμε παρανομίες ή απάτες όσον αφορά, δεν απαγορεύεται δηλαδή κάτι τέτοιο, ωστόσο σε γενικές γραμμές δεν μπορεί να οδηγήσει σε σωστή και βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνονται υπόψη οι ε, συγκεκριμένες, ε, ε, οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ισχύουν για κάθε αγροτική περιφέρεια και να λαμβάνονται οπωσδήποτε υπόψη και τα εθνικά προγράμματα ενέργειας αλλά και τα εθνικά προγράμματα για τις ανανεώσιμες. Επίσης η Κομισιόν θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το ρόλο του ΙΑΡΕΦ ε, και να ζητήσει από τα κράτη-μέλη ε, να δώσουν ε, και να δίνουν γενικότερα συγκεκριμένες πληροφορίες όσον αφορά τα προγράμματα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την υλοποίησή τους για το 2019. Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ένα καλύτερο ξεκαθάρισμα έτσι ώστε να επιλέγονται αυτά τα προγράμματα για τις ανανεώσιμες πηγές που θα έχουν σαν σαν αποτέλεσμα και την ε, σωστή ανάπτυξη της ε, υπαίθρου. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια και είμαι στη διάθεσή σας ε, για οποιοδήποτε διευκρίνηση. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η εισηγήτρια, κύριε Κάντενμπαχ. Ίσως είναι καλό που λείπει η κυρία Γκρέσλε, γιατί πάλι θα εκνευριζότανε. Γιατί έχουμε και εμείς την ίδια κατάσταση. Υπάρχουν κάποιοι στόχοι, τους οποίους έχουμε θέσει ήδη για τον εαυτό μας και το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να αποδείξουμε ότι τα χρήματα δαπανώνται σύμφωνα με το κονδύλι που έχει προγραμματιστεί τις προσδοκίες και τις ελπίδες ξέρουμε ότι αυτό αφορά ένα κλάσμα και μόνο των χρημάτων και αυτό είναι τροφή για σκέψη. Και δεύτερον, τα υπόλοιπα μέσα, τα ακούσαμε τώρα και από το ελεγκτικό συνέδριο με τρόπο δραματικό και τραγικό, ότι σε πολλές άλλες περιπτώσεις δεν είναι σαφής ότι κάνει δείκτες και είναι πολύ δύσκολο για το ελεγκτικό συνέδριο και σε τελική ανάλυση και για το φορολογούμενο να διαπιστώσει εάν και κατά πόσο τα κονδύλια αυτά πραγματικά έρχονται να προσθέσουν την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και στη συγκεκριμένη περίπτωση για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Γιατί πάντα ε, στα γερμανικά υπάρχει μία ε, έκφραση που λέει ότι τα, τα, χρήματα δεν έχουν ε, μέτρο. Ε, εδώ έχουν μέτρο, έχουν και προέλευση και έχουν και συγκεκριμένο προορισμό. Και στην ανακοίνωση του Επιτρόπου Χόγκαν για τη μελλοντική γεωργική πολιτική να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα ελιγμών στα κράτη-μέλη. Και ε, θα ακούσουμε και πάλι από την Επιτροπή αυτά που μας λέει Πάγια, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά, διότι είναι στα χέρια των κρατών μελών. Το πώς θα χειριστούν αυτά τα προγράμματα, πώς θα χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια και πώς θα τα διαμορφώσουν. Κατά την άποψή μου, ε, δεν είναι αυτό ο στόχο των συγκεκριμένων χρημάτων, να αποφασίσουν τα κράτη-μέλη κατά το δοκούν και ε, με τρόπο που είναι δύσκολα εμ, μετρήσιμος και ελέγξιμος. Και θέλω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα ε, λάβει πολύ σοβαρά υπόψη και όχι ελαφρά όπως ακούσαμε για τη μελλοντική ε, γεωργική πολιτική και το μελλοντικό δεύτερο πυλώνα. Να έχουμε αυτήν την ε, στόχευση, τη στήριξη της υπαίθρου. Αυτή τη στιγμή έχουμε την εντύπωση. Εντάξει, είναι σημαντικό να περάσουμε στις ανανεώσιμες, αλλά έχουμε λίγο την εντύπωση ότι είναι μόνο ένα μέσο χρηματοδότησης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και ένα σημείο που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό είναι το θέμα της στήριξης της βιομάζας. Και σε πολλέ άλλε συζητήσει το έχουμε πει και λυπάμαι που δεν έχουμε δώσει συναδέλφου από την Επιτροπή Γεωργία είναι την Επιτροπή Περιβάλλοντο. Και η βιομάζα δεν είναι κάτι ε, το βιώσιμο απαραίτητο. Και θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε και αυτό. Νομίζω ότι πέρασε και ο χρόνος μου. Ελπίζω να έχουμε τις δυνατότητες Γιατί ο κόσμος δεν έχει κατανόηση για τις δαπάνες στο γεωργικό τομέα. Και πρέπει να μιλήσουμε και για το Brexit. και για τη μελλοντική γεωργική πολιτική και μετά το Brexit θα είναι λιγότερα τα χρήματα και θα πρέπει να αναρωτηθούμε πού θα γίνουν οικονομίες και περικοπές. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ο δεύτερος πυλώνας. Είναι πάρα πολύ επιπόλαια και τσαπατσούλικη η ε, ε, ενίσχυση και καθόλου στοχευμένη. Και υπάρχει κίνδυνος να γίνουν οριζόντιες περικοπές και χοντρές, αδρές, έτσι. Αυτό είναι εις βάρος και της ανάπτυξης υπαίθρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαίων πολιτών. Πραγματικά, κοιτάξτε αυτές τις προτάσεις για να μπορέσουμε να αποδεικνύουμε ότι ε, τα χρήματα των φορολογουμένων χρησιμοποιούνται ε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ανταποκρίνονται και στους στόχους μας που έχουμε θέσει είτε είναι για το κλίμα, οτιδήποτε και τους πετυχαίνουμε. Ευχαριστώ. Είναι μια δεύτερη συζήτηση ε, ως συνέχεια της έκθεσης, γι' αυτό θα πάρει λίγο παραπάνω χρόνο. Λοιπόν, συστάζω στον κύριο Σντεχόφσκι το λόγο. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τον έγγραφο και για την προφορική παρουσίαση. Είπατε ότι μάλλον καλό είναι που δεν είναι εδώ η κυρία Γκρέσλε, γιατί θα τα είχε πάρει κρανιογκεφαλικά. Ίσως είστε σε καλύτερη θέση εσείς να είστε η επόμενη πρόεδρος της Επιτροπής μας. Θέλω να ευχαριστήσω τέλος πάντων το ελεγκτικό συνέδριο για να σοβαρευτώ. Είναι μια πολύ καλή έκθεση αυτή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αγροτική ανάπτυξη. Πολλές φορές ε, σας κοίται κριτική και υπάρχουν ειδικέ εκθέσεις για αυτό το θέμα. Αλλά πρόοδο δεν βλέπουμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Πολλά από τα προγράμματα αυτά περιγράφονται αναλυτικά, δεν έχουν όμως δείκτες αξιολόγησης ε, και είναι τελείως τυχαίες ε, δεν υπάρχει καμία συνέπεια στην προσέγγιση. ανανόσιμε πηγές ενέργεια καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα. Αφορούν το κλίμα, συνολικά όλα αυτά θα επηρεάζουν γενιές και γενιές. Δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό, αλλά θα εξαρτηθεί από το τι εμείς θα αποφασίσουμε σήμερα, από τις επιλογές που θα κάνουμε εμείς σήμερα. Είναι στην πρώτη γραμμή για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων η Ένωση στον κόσμο. Έχει τεράστιες φιλοδοξίες για την επίλυση αυτών των προβλημάτων και είναι θετικό που είμαστε τόσο φιλόδοξοι. Όμως είναι σημαντικό, δεν είμαι ο πρώτος που το λέω άλλωστε, να μην χαθεί έτσι το δυναμικό της Ένωσης, να μην ε, εκπνεύσει τόσο απλά, τόσο εύκολα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να φροντίσει όλα τα κράτη-μέλη να κάνουν τα δέοντα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι σημαντικές για την ασφάλεια αφοδιασμού, αλλά και από γεωπολιτικές πλευράς. Έχουν σημασία για την ανεξαρτησία μας, την ενεργική μας αυτονομία ενέργεια από πηγέ, πηγές, αγροτική ανάπτυξη. Πολύ ενδιαφέρουσα διασύνδεση των δύο. Θέλουμε αλλαγέ. Ε, να έχει φωνή η περιφέρεια, γιατί εκεί μπορούν να προωθηθούν καλά project και για την βιοενέργεια. Συμφωνώ με το ελεγκτικό συνέδριο και τα πορίσματά του μπορούν να υπάρξουν συνέργειες στο πεδίο αυτό. Είναι τεράστια τα περιθώρια. Και είναι λυπηρό. Πολύ λυπηρό που το ελεγκτικό συνέδριο θεωρεί ότι δεν μπορούν να επιτευχθούν όμως οι συνέργειες αυτές. Είχαμε την ειδική έκθεση 31 το 2016 που λέει ότι ένα πέμπτο του προπολογισμού της Ένωσης πρέπει να δαπανηθεί για δράση στον τομέα του κλίματος και πρέπει η Κομισιόν να εκπονήσει ένα στρατηγικό σχέδιο για τον προπολογισμό, για μέτρα για το κλίμα. Απευθύνω έκκληση στην Κομισιόν. Γεωργία, αλία, αγροτική ανάπτυξη. Πρέπει αυτά τα θέματα να είναι στο επίκεντρο σε σχέση με την κλιματική περιβαλλοντική πολιτική. Αυτά από το 16, τα έλεγε το Ευρωπαϊκό Συνέδριο, και είμαστε στο 18 και δεν έχει γίνει τίποτα. Θέλω συγκεκριμένη, συγκεκριμένη και ξανά ματά, μανά, συγκεκριμένη στρατηγική από την Κομισιόν για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να λαμβάνει υπόψη όλες τις δυνατικές πτυχές ε, του Ενωσιακού προπολογισμού και τη διασύνδεσή τους. Να μην ε, κάνουμε στεγανοποίηση και χωρίζουμε τα θέματα σε κατηγορίες. Το θέμα να προωθήσουμε προσθέμενη αξία. Δεν τα ακούτε για πρώτη φορά, αλλά είναι σημαντικά αυτά που λέω. Τα έργα, τα σχέδια θα πρέπει να βασίζονται σε, μια, σε έναν σε βάθος προβληματισμό που θα έχει θέμα. Το γιατί ε, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θέλουμε να πετύχουμε. Έρχεται το Παρίσι στο μυαλό μας για τα κλιματικά. Και βέβαια η Κομισιόν πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν συνέργειες, πραγματικές, τοπικές στρατηγικές. Θα σχετίζονται βέβαια και με τον νησιακό επίπεδο, γιατί τέλος δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Και κλείνω λέγοντας, ναι είναι πρόκληση. Οι προκλήσεις μου αρέσουν πολύ όμως εμένα. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις αυτές και Πιστεύω στο μέλλον θα έχουμε συγκεκριμένα αυτά αποτελέσματα και δεν θα ασκούμε πλέον κριτική, αλλά θα δίνουμε επένους στην Κομισιό. Πρόεδρος. Ο επόμενος που θα τα πάρει με το θέμα αυτό φαντάζομαι είναι ο κύριος Λάναγκαν. Ευχαριστώ πολύ. Σωστά είπατε ότι δεν ε, υπήρχε μεγάλη διασύνδεση με, τις, ε, ε, με την Ήπεθρο και ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ναι, αλλά ποιος άλλος έπρεπε να ληφθεί υπόψη αφού περί της Ήπεθρου πρόκειται. Ε, λέτε για βιώσιμη, λέτε ότι υπάρχει μεγάλο δυναμικό και για συνέργειες ε, και για ανάπτυξη της υπαίθρου. Πρέπει να σας πω ότι στη δικιά μου περιφέρεια ε, υπάρχουν πολλά προγράμματα για τις ανανεώσιμες πηγές, αλλά καμία μηδέν, μηδενική διασύνδεση με τον τοπικό πληθυσμό και με την τοπική κοινωνία. Ε, κοιτάξτε, εμείς ε, ζούμε σε μια περιοχή ε, όπου με την τύρφη που βγάζουμε από το χώμα κάνουμε τα πάντα. Ζεσταίνουμε τα σπίτια μας, τα, στεγνώνουμε τα ρούχα μας. Μιλάμε για ε, ε, πληθυσμούς, μιλάμε για περιοχές οι οποίες θα πρέπει να μετακινηθούν προς νέες λύσεις και αυτό είναι εξαιρετικό. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι όχι μόνο ε, δεν προκύπτουν συνέργειες, αλλά ενώ είχαμε μία ανεξαρτησία λόγω της τύρφης, την οποία όμως δεν μπορούσαμε να την... δεν ήταν ιδιοκτησία μας και δεν είχαμε την πλήρη η εξουσία ας πούμε ε, ε, πάνω στο θέμα αυτό ενδεχομένως, ενδεχομένως θα βρεθούμε σε μια κατάσταση που θα είναι πολύ χειρότερα γιατί ναι μπορεί να ε, ε, θέλουμε να έχουμε κάποιες, ε, κάποια επιστροφή όσον αφορά αυτή η χρήση αυτών των νέων ενεργειών αλλά για την ώρα δεν έχουμε τίποτα και επίσης όσον αφορά αυτό το τεράστιο θέμα της βιομάζας υπάρχουν ντόπιοι πληθυσμοί οι οποίοι δεν ασχολούνται καθόλου, δεν, δεν εμπλέκονται καθόλου με το θέμα, ούτε καν αυτοί που ασχολούνται με την υλοτομία. Εμείς ε, ε, ε, έχουμε δει πολλές περιπτώσεις όπου έχουμε κάποιες γεές οι οποίες έχουν καλλιεργηθεί με συγκεκριμένα ε, με συγκεκριμένους ε, σπόρους ε, για παραγωγή βιομάζας και στην ουσία έχουμε ήδη παράγει πάρα πολλούς ρήπους, πάρα πολλές εκπομπές και από τη μία λέμε ότι κάνουμε προσπάθειες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από την άλλη μεριά τελικά μέσα από αυτές τις καλλιέργειες δημιουργούμε, προκαλούμε περισσότερες εκπομπές, περισσότερες περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα από ότι με τις μέρες Δεν χρειάζεται να κάνεις κανεί ιδιοφυή έτσι ώστε να καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά με όλα αυτά εγώ προέρχομαι από μια περιοχή όπου έχουμε ανεξαρτησία όσον αφορά ε, το, το, το, καύσιμο. Ακόμα και όταν είμαστε πάμπτωχοι και δεν είχαμε να φάμε, ε, πραγματικά είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε ε, ένα καύσιμο. Τώρα είμαστε ακόμα σε ακόμα χειρότερη κατάσταση και νομίζω ότι όλη αυτή η διαδικασία στην ουσία δεν προωθεί την πρόοδο και έχετε δίκιο. Πρέπει να ξέρουμε τι κάνει και η Κομισιόν επιτέλους. Ε, και ε, όσον αφορά τη βιομάζα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι δυνατόν να καταστρέφουμε πρωτογενή παραγωγή για να παράγουμε ε, βιομάζα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε ακριβώς πώς έχει η κατάσταση. Θα πρέπει να δούμε την, το σύνολο της διαδικασίας. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι ο άνθρακας όταν καίγεται παράγει ρήπους και όταν καίγεται η βιομάζα να μην βλέπουμε τους ρήπους που παράγει και τη μόλυνση. Ευχαριστώ. Τώρα να ακούσουμε τι σκέφτεται για όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Χόφμαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ο κύριο καλά δεν πειράζει. Χόφμαν πάντως είμαι. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρία Κάντεμπαχ, κύριε Γέρεπ. Θέλω να πω στην εισηγήτρια και στο ελεγκτικό συνέδριο ευθύ εξ αρχή, Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις εκθέσεις. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσε και για μας, γιατί δείχνουν κάποια σημεία όπου υπάρχει χώρος για βελτίωση, για να το πω έτσι, όπως είπατε και εσεί προηγουμένως. σε ό,τι αφορά το μέλλον της πολιτικής για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υπάρχει νομοθετική πρόταση επιτάπητος, την οποία συζητάει και το Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή και κάποια στοιχεία που θα μας ε, βοηθήσουν να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ορισμένα από τα σημεία που αναφέρατε κι εσείς. Um, και ιδιαίτερα το, το θέμα είναι ότι χρειάζεται να ε, αυξηθεί το κριτήριο βιωσιμότητας της βιοενέργειας of που σημαίνει η χρήση της βιομάζας και της παραγόμενης ενέργειας με κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες για τη χρήση βιομάζας από δάση. Να έχουμε ένα πώς να το πω, ε, επίπεδο με αντίστοιχη κατάσταση για να μπορούμε να κρίνουμε Αναφερθήκατε σε μερικά σημεία που θέλετε στο μέλλον να βελτιωθούν, γιατί μας είπατε ότι δεν έχετε ενημέρωση και πληροφορία για να μετρήσετε τι κάνει και τι δεν κάνει η ε, πολιτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου, την αγροτική ανάπτυξη. Αν μου επιτρέπετε να απαντήσω σε ένα σημείο. Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο μετρούμε ε, ως δείκτες αποτελεσμάτων τη δράση υποστηρίξη δραστηριοτήτων στο συγκεκριμένο τομέα. Οι δείκτες αποτελεσμάτων ε, δεν ε, είναι κάτι που μπορεί να μετρηθεί κάθε χρόνο. Θα έχουμε λοιπόν τα αποτελέσματα το 2019 με ειδική έκθεση αντίστοιχα και με πληροφόρηση για το σύνολο των επενδύσεων στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και θα έχουμε και ένα δεύτερο δείκτη την ανανεώσιμη ενέργεια που έχει παραχθεί από επιδοτούμενα έργα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί έχουμε μετρήσιμους δείκτες. Και σας διαβεβαιώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αγωνιά να έχουμε δείκτες, αλλά το πρόβλημα είναι ότι τα κράτη-μέλη αντιδρούν. Για να είμαι ειλικρινής, για την πολιτική της αγροτικής ανάπτυξης έχουμε ένα κοινό σύστημα και πλαίσιο ελέγχου και αξιολόγησης, όπου έχουμε ορίσει δείκτες που πρέπει να μετρούν τα κράτη-μέλη, οφείλουν να το κάνουν, ε, και σε πολλούς τομείς, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να είναι αναλογικά με τις προσπάθειες που κάνουν και τα κράτη-μέλη. Και δεν είναι πάντα εύκολο να εντοπίσει κανείς σε ένα συγκεκριμένο έργο την ποσότητα ανανεώσιμης ενέργειας, ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Ξέρουμε ότι είναι σημαντικό αυτό, το προχωρούμε. Το 2019 θα υπάρξει κάποια σχετική πληροφόρηση. Ε, για το μέλλον τώρα και το μέλλον ε, νομοθετικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Μπορεί να γνωρίζετε από την ανακοίνωση για το μέλλον της γεωργίας και των τροφίμων ότι ε, προτιθέμεθα να προβούμε σε κάποιες βελτιώσεις. Μία από τις βελτιώσεις αυτές είναι σαφέστατα η ιδέα ότι θα βασίζουμε την πολιτική μας στα αποτελέσματα και στις επιδόσεις, να δούμε τι βγαίνει από την εκάστοτε πολιτική. Όχι τι έχουν κάνει τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, αντιστρέφουμε τη θεώρησή μας. Επίσης θα ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να κάνουν πολύ ειλικρινή ανάλυση των τοπικών αναγκών σε κάθε έργο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Των τοπικών αναγκών. Δεν αφήνουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν ό,τι θέλουν ή ό,τι θα προτιμούσαν. Αλλά τι χρειάζονται οι περιφέρειες και τα κράτη-μέλη. Δεν χρειάζονται όλοι τα ίδια πράγματα και θα πρέπει να τους επιτρέψουμε να βασίσουν τις ιδέες και τη στρατηγική τους σε μια επιτόπια ανάλυση, χωρίς να τους επιβάλλουμε μια ιδέα παντού σε όλα τα κράτη-μέλη για το τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να ενισχύσουμε αυτού του είδους λοιπόν την ανάλυση. επίσης και σε αυτό που προτείνεται για ένα εργαλείο ελέγχου γενικό, ένα εργαλείο αξιολόγησης για όλες τις υπόλοιπες πολιτικές. Δηλαδή όλες οι υπόλοιπες πολιτικές πώς επιδρούν στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Στο μέλλον θα έχουμε κοινούς δείκτες, όπως και τώρα, και θα μετρούμε επίσης και ε, στόχους της ανανεώσιμες. Υπήρξε μια ιδέα να καθοδηγούμε περισσότερο να βοηθούμε τα κράτη-μέλη. Είπε και ο κύριος Φλάναγαν ότι στη δική του περιφέρεια δεν υπάρχουν τέτοια έργα ε, στον πληθυσμό. Έχουμε ειδική αναφορά και έκθεση για τα έργα που έχουμε στην ανάπτυξη πέθουμε ξεχωριστή στο σελίδα ε, και στις ανανεώσιμες, ακριβώς εκεί έχουμε βάλει παραδείγματα. Δεν είναι μόνο τα φωτοβολταϊκά ή ε, οι που και αυτά τα υποστηρίζουμε, αλλά ε, είναι ε, τοπικές πρωτοβουλίες, έχουμε και παραδείγματα που το δείχνουν και μια εταιρική σχέση για την καινοτομία με συγκεκριμένη εστιασμένη προσπάθεια και ομάδα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με βέλτιστες πρακτικές. Δηλαδή γίνονται πολλά πιστεύω έτσι ώστε να ενημερώνονται τα κράτη-μέλη για τις δυνατότητες που υπάρχουν και τις ευκαιρίες. Ελπίζουμε να ε, το ακολουθήσουν και να το υιοθετήσουν σε μεγάλο βαθμό αυτά τα κράτη-μέλη. Και επίσης στο μέλλον θα υποχρεώσουμε να επιβάλλουν ε, κριτήρια επιλογής, ε, επιλεξιμότητας δηλαδή για την επιλογή των προγραμμάτων και των έργων και να υπάρχει και μια κοινή μεθοδολογία έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα πιο ποιοτικά προγράμματα και έργα θα επιλέγονται. Ευχαριστώ πολύ. you, Ευχαριστώ. Θα δώσω τη δυνατότητα στο ελληνικό συνέδριο να απαντήσει σε οτιδήποτε θεωρεί σημαντικό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω για τις απόψεις και την υποστήριξη στα πορίσματά μας. Να δώσω κάποιες απαντήσεις στον κύριο Φλάναγκαν. Συμφωνώ με όσα είπατε 100%. Μίλησα αρχικά για τα ζητήματα βιωσιμότητας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι συνώνυμες με βιώσιμότητα. Δεν είναι πάντοτε βιώσιμες οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα πρέπει λοιπόν ε, να προσέχουμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τη βιομάζα. Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις ανώσιμες πηγές ενέργειας. Μιλάγατε για μεγάλα έργα, αν κατάλαβα καλά. Οι ανανόσιμε πηγές ενέργειας χρηματοδοτούνται από πολλά διαφορετικά ταμεία, είπαμε. Αλλά εμείς εστιάσαμε σε ένα μόνο, στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και όχι ε, άλλες επενδύσεις ε, και άλλες ε, μονάδες εγκαταστάσεις. Σε ό,τι αφορά το τι λάβαμε υπόψη, αν όχι τι αγροτικέ περιοχές. Εμείς, ειδικώ για αυτό το ταμείο αγροτική ανάπτυξη, θέλαμε να δούμε πώς σχεδιάζουν τα κράτη-μέλη τι δαπάνε των κονδυλίων αυτού του ταμείου και πώς σχετίζουν τις επενδύσεις ανανεώσιμε πήγες με την ανάπτυξη της υπαίθρου. Και εξήγηση δεν βρήκαμε ή μάλλον σχέση δεν βρήκαμε Γι' αυτό και λέμε στην έκθεσή μας ότι κάποιε επενδύσεις έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αγροτική ανάπτυξη από ό,τι άλλες. Αν έχετε έναν αγρότη που βάζει φωτοβολταϊκά ε, στην οροφή ε, της ε, φάρμας του για δική του χρήση, δεν βοηθάει και τόσο αυτή την αγροτική ανάπτυξη. Αλλά αν χρηματοδοτεί κάποιο την παραγωγή της, του δικτύου θέρμανσης και χρησιμοποιεί τα πέλετς ή κάτι άλλο, δημιουργεί μια λυσίδα ε, εφοδιασμού. Για την προετοιμασία των ε, κομματιών αυτοξύλου που χρησιμοποιούνται για, το... για τη θέρμανση, απασχολούνται περισσότεροι άνθρωποι κτλ. Το θέμα είναι τι κάνουν τα κράτη-μέλη με αυτά τα χρήματα. Και ένα ακόμη σχόλιο σε σχέση με αυτό που είπε η κυρία Λούρις Χόφμαν από την Επιτροπή, είπατε για το 2019 ότι τότε θα έχετε κάποιους δείκτες για τα αποτελέσματα, για το ποιε θα είναι οι συνολικές επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργεια. Αυτό είναι πιο πολύ ε, για το output και όχι για τα αποτελέσματα. Ε, και σίγουρα το δεύτερο που είπατε ε, θα βελτιώσει την κατάσταση, αλλά αν, μας, ε, αν παρακολουθήσετε μόνο έναν δείκτη αυτόν που είπατε, δηλαδή ε, ποσότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τότε ένα μόνο πρέπει να το ταμείο που θα αντιχρηματοδοτεί την ανανεώσιμη ενέργεια. Η χρηματοδότηση μέσω του Γεωργικού Ταμείου Χρωτικής Ανάπτυξης σχετιζόταν με την ανάπτυξη της υπαίθρου. Αλλά θέλουμε δείκτες. Τι δημιουργήθηκε, δημιουργήθηκε με τι επενδύσει απασχόληση, δουλειέ, κάτι άλλο. Όχι μόνο παραγωγή ανανεώσιμη ενέργεια. Πρέπει να καλύπτονται και άλλα θέματα. Ευχαριστώ τέλο η συγγήτρια. Το ερώτημά μου κατακλείδει προς την, αντίστοιχη, προς την ίδια κατεύθυνση πηγαίνει, δηλαδή με αυτούς τους δείκτες. Το 2019 λέτε. Δεν είναι και τόσο ευτυχής επιλογή, γιατί ε, θα έχουμε τις επόμενες εβδομάδες ε, ε, συγκεκριμένη νομοθετική πρωτα... πρόταση από την Κομισιόν για την κοινή πολιτική. Και νομίζω ότι είναι ατυχές να περιμένουμε χρόνια για να δούμε πώς θα δημορφωθεί ο δεύτερος πυλώνας και το δεύτερο σε ό,τι αφορά αυτό το σύνδεσμο μεταξύ ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των επιπτώσεων που έχει στις ε, περιφέρειες. Πώς θα το μετρήσουμε αυτό. Ε, δεν πρέπει να υπάρχουν κάποιες λίστες ιεράρχησης ε, για τα προγράμματα των κρατών μελών. Πώς θα τα μετρήσουμε και θα τα εξολογήσουμε Δεν θα έχουμε διάλογο, γιατί έχουμε μείνει 15 λεπτά πίσω. Κακός, λέει κύριε Κάτι. Εντάξει, τότε σταματώ εδώ. Ευχαριστώ. Ένα ακόμα ενδιαφέρον θέμα και άλλη μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είπε κανεί ότι είναι βαρετή η Επιτροπή μα Και το επόμενο θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον. Πάμε στο 9 ξανά, γνωμοδότηση για την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξη για το πώ θα επηρεάσει η πολιτική συνοχή στη Βόρεια Ιρλανδία. Ενδιαφέρον το θέμα, γιατί εγώ γνωμοδοτώ για την έκθεσή μου εδώ πέρα. Λίγο ασυνήθιστο και δεν ήξερα και κατά πόσον επιτρέπεται κάτι τέτοιο, αλλά μου είπαν σίγουρα θέλετε το λόγο κύριε Φλάραγκαν, ήμουν βέβαιος γι' αυτό. Λοιπόν, είχαμε να κάνουμε αυτή την ε, γνωμοδότηση, έχετε, ε, σας έχει μοιραστεί, μάλλον έχετε στο φάκελό σας και ένα αντίγραφο αυτής της ε, γνωμοδότησης. Εγώ βέβαια προσπάθησα να δω τα κεντρικά στοιχεία ε, όσον αφορά το κοινωνικό ταμείο δηλαδή και το ε, ERDF ε, και το ΕΤΠΑ ε, και την στρατηγική μετά το 2020. Ε, Επίσης ε, έκανα και μία επίσκεψη σχετική με την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Είδαμε από κοντά κάποια προγράμματα διασυνοριακά που δίνουν την δυνατότητα να διευκολύνονται αυτοί που ζουν στη μία πλευρά των συνόρων και εργάζονται στην άλλη. Ε, καθώς επίσης ε, και ε, προγράμματα τα οποία βοηθούν την διασυνοριακή παροχή υγείας. Επίσης είδαμε από κοντά και μελετήσαμε και κάποια προγράμματα ειρηνευτικής διαδικασίας σχετικά ας πούμε με την υπηρεσία των επιζώντων και των θυμάτων. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Επίσης επισκεφθήκαμε κάποια κοινοτικά κέντρα ε, σε διάφορες ε, περιοχές, ε, δύο συγκεκριμένα, συνδέονται δε με αυτά τα κοινοτικά κέντρα και κάποια προγράμματα συνένωσης και συμβίωσης όπου οι άνθρωποι παίζουν ποδόσφαιρο μαζί, κάνουν, χορεύουν μαζί και τα λοιπά και αυτό νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ συγκλονιστικό. Είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι μετά από πολλά χρόνια ξαναβρίσκονται βρίσκονται αντιπαράθεσης και ε, προβλημάτων, ξαναβρίσκονται κοντά και κάνουν ε, μαζί διάφορα πράγματα. Ε, αυτά είναι προγράμματα Interreg και προγράμματα τα οποία εντάσσονται στην διαδικασία ειρήνευσης και αυτό είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουν και μετά από το Brexit. Θα πρέπει να πείσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά βεβαίω και τις άλλες δύο πλευρές, ε, την ε, Ιρλανδική κυβέρνηση και την Βρετανική κυβέρνηση ε, γιατί πραγματικά η επίπτωση στι δύο κοινότητε τέτοιων προγραμμάτων και τέτοιων σχεδίων είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να συνεχίσει και μετά το Brexit. Επίσης μου είχαν πει πριν πάω κιόλας ότι θα έπρεπε να κρατήσω το στόμα μου κλειστό όσον αφορά τον Brexit όσο ήμουν εκεί. Δεν είναι και πολύ εύκολο βέβαια κάτι τέτοιο γιατί η συζήτηση πάντα στρέφεται για την περίοδο μετά το 19 ε, και βεβαίω το μεγάλο, το κεντρικό ζήτημα είναι το θέμα των συνόρων, του συνόρου μάλλον και ε, αυτά δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ε, Φαντάζομαι και ελπίζω ότι τα σημεία τα οποία αναφέρω θα βρουν σύμφωνους ε, τους συναδέλφους. Ο κύριος Ζέλερ και μετά ο κύριος Φλάναγκαν. Ευχαριστώ Ντέρεκ. Είχα την τιμή εγώ να προεδρεύω στην Διερευνητική Επιτροπή της ε, ε, αποστολή μάλλον της Επιτροπής περιφερειακής ανάπτυξης στη Βόρεια Ιρλανδία. Και αν θέλει κάποιος να δει τόπο τα ευρωπαϊκά προγράμματα και να πιστεί που έχουν αποδειχθεί στην πράξη, να πάει στη Βόρεια Ιρλανδία. Καμιά φορά στις ειδήσει αυτά περνάνε στα ψηλά. Θυμάστε τις ειδήσει πριν από 25 χρόνια. Δεν περνούσε μέρα σχεδόν που να μην είχαμε βόμβες, βία επεισόδια στη Βόρεια Ιρλανδία. Είτε αυτό ήταν στο Μπέλφαστ είτε στο Ντέρι. Σήμερα ούτε καν το νιώθει κανείς αυτό. Πολλοί μας είπαν όμως να μην σας γελάει η επιφάνεια. Εμείς το οφείλουμε αυτό στο γεγονό ότι είμαστε μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν υπάρχει αίσθηση συνόρων. Πηγαίνω έρχεται ο κόσμος από τη Βόρεια Ιρλανδία στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας χωρίς προβλήματα και με δισεκατομμύρια έχει χρηματοδοτήσει εδώ τα προγράμματα Ευρωπαϊκή Ένωση που πραγματικά σέφεραν στην ειρηνική συμβίωση. Εάν δεν υπήρχε κάτι τέτοιο δεν έχει καμία εγγύηση κανείς να δώσει ότι θα συνέβαινε ή ότι θα συμβεί στο μέλλον κάτι τέτοιο. Ο Μπράιν Χέις, εκλεκτός Ιρλανδός συνάδελφος και ο με παρακάλεσε να πω δύο λόγια για τη γνωμοδότηση του Ντέρεκ Βον και θα σας διαβάσω αυτό το σκονάκι που μου έχει δώσει, με χαρά. Γράφει λοιπόν ο Brian Hayes ε, στα αγγλικά. Χαιρετίζω και ε, καλωσορίζω την γνωμοδότηση του Derek Vaughan. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τις ευεργετικές επιπτώσεις στη Βόρεια Ιρλανδία. Τα προγράμματα Peace, Interreg και η Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση είχαν πολύ θετικό αντίκτυπο. Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο του PDP ε, η Βόρεια Ιρλανδία και οι ε, παραμεθόριες κομιτείες ε, πάρουν πάνω από 500.000 ευρώ. Αλλιώς δεν θα είχαν υλοποιηθεί πολλά σημαντικά έργα. Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα στον Τέρι και στον Τάναγκαλ, εκατέρωθεν των συνόρων, προωθεί την αταλλαγή επιχειρηματιών στην περιοχή. Άλλο έργο, συνεργασία και αφορά την κοινωνική ανάπτυξη και θέματα δημόσιας υγείας, ε, πρόληψη της παχυσαρκίας, υποστήριξη παιδιών ε, αυτιστικών. Χωρίς την υποστήριξη λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα υπήρχαν τα περισσότερα προγράμματα αυτά. Καλωσορίζω το γεγονός ότι αναγνωρίζει ο εισηγητής πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά και θαρρύνει τη συνέχιση της χρηματοδότησης συμπέρασμα. Δεν αφιβάλλει κανείς ότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχή είχε ευεργετικές ε, Επιπτώσει στη Βόρεια Ελλαδία. Καλωσορίζω τη γνωμοδότηση, ε, ε, αυτά που λέει ο εισηγητή για τη λύση μετά το 2020. Όλα αυτά τα λέει ο κύριος Χέις. Ευχαριστώ που το αναγνώσατε. Ο κύριος Φλάναγκαν. Και ε, εγώ με τον Brian Hayes διαφωνώ σε πολλά πράγματα, αλλά όχι σε αυτό που μόλις ακούσαμε. Συμφωνώ 100%. Και σας ακούω να μιλάτε για κατάσταση πριν από 25 χρόνια άνοιγε τη τηλεόραση και άκουγες για κάποια καταστροφή που έγινε. Και πάντα θυμάμαι κάτι που είχε πει ε, ο φίλος μου, Σον Ρίγκαν, που δυστυχώς δεν είναι μαζί μας. Πριν από τρία χρόνια μου είπε τώρα θα πάω στον τέρι και μπορώ να καθίσω με την πλάτη στη βιτρίνα ή σε παράθυρο χωρίς να φοβάμαι ότι θα με πυροβολήσουν ή ότι θα μου συμβεί κάτι. Είναι πραγματικά ανατριχιαστικό αυτό και η έκθεσή σα, Ντέρεκ, είναι εξαιρετική. Χρειαζόμαστε το πρόγραμμα Interreg και τη χρηματοδότηση του ερμηνευτικού προγράμματο. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συνεχιστεί αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχει αποδώσει και υπάρχει μια παράνοια κάπου ότι τα χρήματα δεν τη χάνουν καλής διαχείρισης. Ε, μέχρι και τελευταία δεκάρας είναι το αυτό και μέχρι το τελευταίο σέντ του, του λεπτού. Και από πλευρά ελέγχου του προπολογισμού μην ανησυχείτε, γιατί γι' αυτό μιλάμε. Πιάνουν τόπο τα χρήματα και πάρα πολύ μεγάλο και στο παρελθόν και στο μέλλον θα συνεχιστεί αυτό. Αποφύγατε να αναφερθείτε στο Brexit, αλλά στην έκθεση, στο σημείο 3, λέει κάτι πολύ σημαντικό ε, δεν μπορούμε να δούμε ποια ε, λύση θα βρεθεί για τη Βόρεια Ελλάδα μετά το 2020. Προσοχή, ε, στο Ιρλανδικό Κοινοβούλιο υπήρξε ένα ενιαίο μέτωπο διακομματικό ότι οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά. Τώρα όμως υπάρχει αίσθηση ότι καθώς προχωρούν οι συνομιλίες για το εμπόριο χωρίς να αποφασίσουν ουσιαστικά τι θα γίνει με τα σύνορα, Έχουμε οδηγηθεί σε μια κατάσταση όπου το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα στη Βουλή που υποστηρίζει και την κυβέρνηση τώρα αρχίζει να επικρίνει τη διαδικασία και τις συνομιλίες και το δρόμο που έχουν πάρει. Προσοχή λοιπόν να μην μας ξεφύγει αυτό και να μην μείνουμε πίσω. Μέχρι τώρα καλά τα πήγαμε, αλλά θέλουμε να συνεχίσουμε με την υποστήριξη που παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλή έκθεση λοιπόν. Και πραγματικά για κάποιον που δεν είναι Ιρλανδός, πολύ ε, διάνα πετύχατε. Μα εγώ πάντα χαίρομαι να πηγαίνω, βλέπω και τους καδέλφου μου, τους Κέλτες. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυρία Γκονσάλης Ενάντε. Yes, thank you. Uh, thank you, Chair. Ευχαριστώ. Χαιρετίζετε την έκθεση κομισιών, την γνωμοδότηση. Επίση, χαιρόμαστε που είχατε μια επιτυχή επίσκεψη και είδατε όλα τα καταπληκτικά πράγματα που έχει πετύχει η πολιτική συνοχή πράγματι στην Βόρεια Ιρλανδία. Θεωρούμε και εμεί ότι είναι θετικό ο αντίκτυπο πολιτική αυτή. Ένα σημείο θέλω να σχολιάσω. Έγινε λόγο για το πρόγραμμα PEACE στην έκθεση και στην γνωμοδότηση και αναφέρεται ω πρόγραμμα για τη Βόρεια Ιρλανδία. Όμω δεν καλύπτει μόνο τη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά την Ιρλανδία εν γέννη. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς αναφέρουμε. Ή θα αναφέρουμε και τα δύο κράτη δύο περιοχές ή θα μιλήσουμε για το πρόγραμμα Peace. Ίσως είναι πιο εύκολο αυτό. Επίσης καλωσορίζουμε την άποψή σας ότι πρέπει να συνεχίσει η διασυνοριακή αυτή ε, συνεργασία παρά την ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2017, όπου είχαμε ήδη πει ότι είμαστε υπέρ να παραμείνουν οι διαχειριστικές δομές, δεν ξέρω τι ε, προβλέπετε. Και περιμένω αύριο και τι θα γίνει στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Δεν έχω πολλά να πω, αλλά σημαίνω αυτό που είπατε ότι καλύπτει και τις δύο χώρες, και την Ελλαδία και την Βορλανδία και ε, έχετε πολύ δίκιο κι εσείς ε, και οι διαπραγματεύσεις για το Brexit. Βέβαια δεν μίλησα εγώ ε, ακριβώς γι' αυτό ε, στην εκθεσή μου, αλλά σίγουρα είναι πολύ καθοριστικός παράγοντας και για το σύνορο Τελωνιακή Ένωση Ενιαία Αγορά. Αν παραμέναμε θα λύνονταν τα προβλήματα. Αυτό το δεν θέλω βέβαια να μιλήσω για το Brexit. Στην επίσκεψη τώρα δεν ακούσαμε κάποια παράπονα, ούτε καταγγελίες για τη δαπάνη των κονδυλίων, φαίνεται ότι έγινε σωστά. Πρέπει να πω ότι τα ε, χρήματα ε, τα δέχονταν γιατί τα θεωρούσαν ουδέτερα, όχι ότι έρχονται από κάποια χώρα συγκεκριμένη. Ε, οι κοινότητες δηλαδή ε, τα ε, αξιοποίησαν τα κονδύλια αυτά γιατί θεωρούσαν ότι προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν επιτυχημένα τα προγράμματα που υποστηρίχθηκαν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να συνεχιστούν ανεξάρτητα του τι θα γίνει το 2019. Για την κατάσταση των απολογιών έχουμε ημερομηνία. Ναι. 30 Απριλίου. Και περιμένω και τις τροπολογίες των συναδέλφων. Εδώ ολοκληρώνουμε και με αυτό το σημείο. Έκλεισε το μικρόφωνο του Πρόεδρου. Η Μαρτίνα που είναι για το τελευταίο θέμα. Α, είναι καθοδόν. Ε, λίγα λεπτά διάλειμμα. Uh, λοιπόν, ήρθε η Μαρτίνα, Επομένω μπορούμε να αρχίσουμε την εξέταση του σημείου 10. Ε, Πρόκειται για ε, θέμα το οποίο αφορά τη συμβολή στην απλούστευση ε, των, του, του προγράμματος έρευνας Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το Horizon 2020. Έχουμε και τον κύριο Μπρένινγκ Μάγερ ο οποίος είναι υπεύθυνο από τη μεριά του ελεγκτικού συνεδρίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, μέλη αξιότιμα της Επιτροπής, ε, κυρίες ε, και κύριοι που ενδεχομένως ακούτε αυτήν την συζήτηση μέσω του διαδικτύου. Θα αναφερθώ στην στο πρόγραμμα έρευνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε μια καινούργια προσέγγιση όσον αφορά του συμμετέχοντε στα προγράμματα έρευνα. Το πρόγραμμα έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, το ισχύον δηλαδή ορίζον 2020, είναι περίπλοκο. 130.000 ε, ε, υποβολές ε, μέχρι τώρα, 20.000 projects τα οποία έχουν λάβει χρηματοδότηση. Πρόκειται λοιπόν για μια περίπλοκη μηχανή η οποία πρέπει παρόλα αυτά να δουλεύει με τρόπο αποτελεσματικό και σωστό. Οι παρατηρήσεις μου από πλευράς του ελεγκτικού συνεδρίου όσον αφορά το πρόγραμμα αυτό είναι ότι μια απλούστευση τέτοιου προγράμματος δεν είναι καθόλου απλή δουλειά. Ε, αυτή, αυτό είναι το κεντρικό μου, ή αν θέλετε, ε, το, το εναρκτήριο σημείο της ε, παρέμβασής μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μετά από τις αλλαγές και τις απλουστεύσεις ενός προγράμματος όπως το Horizon 2020 να είναι ισορροπημένο ανάμεσα σε πολύ ε, διαφορετικά ε, στοιχεία, τα οποία όμως είναι εξίσου σημαντικά ε, όσον αφορά την έρευνα επίσης. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι πρέπει να είναι βαθμιαία η προσέγγιση και η τροποποίηση. Το ελεγκτικό συνέδριο ανέλαβε και την παρουσίαση και την παρατήρηση του προγράμματο Horizon 2020 με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που ε, έδωσε όλα τα απαραίτητα ε, στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν το, τη μελέτη του ενδεχόμενου πλούστευσης αυτού του προγράμματος. Ε, επίσης ζητήθηκε το ενημερωτικό σημείωμα να είναι έτοιμο πριν από τον Απρίλιο έτσι ώστε να ε, ληφθεί υπόψη στον επόμενο προγραμματισμό. Ε, όντως ε, εμείς ε, θα ολοκληρώσουμε ε, και τον Δεκέμβριο μια πιο ολοκληρωμένη έρευνα όσον αφορά την καινοτομία και την έρευνα και εκεί θα αναφερθούν και διάφοροι τρόποι που θα αφορούν τον τρόπο με τον οποίο οι δικαιούχοι βλέπουν και κρίνουν το πρόγραμμα Horizon 2020 η τροποποίηση από πλευρά ε, του Συμβουλίου και της Κομισιόν ε, ε σήμαινε ότι η υπόλοιποι ήταν πάρα πολύ ε, λίγη και επομένως έπρεπε να ετοιμάσουμε πάρα πολύ γρήγορα το έγγραφο βασιζόμενοι σε παλαιότερα έγγραφα του, του, του ελεγκτικού συνεδρίου. Ένα στοιχείο το οποίο είναι απαραίτητο και σημαντικό για τη διαδικασία απλούστευσης ε, είναι το σύστημα ε, των ε, προγραμμάτων και της επιστροφής των χρημάτων. Βλέπουμε ότι τα συστήματα ε, επιστροφής ε, και αποζημίωσης των ε, δαπανών είναι περίπλοκα και πολύ συχνά γίνονται, προβλήματα γίνονται λάθη λόγω και ελλειπούς κατανόησης. Θα είμαι σύντομος γιατί ήδη μπορώ να ξεκινήσω με τα πέντε διλήμματα τα οποία επηρεάζουν την απλούστευση. Το πρώτο είναι απλό. Πολλοί εμπλέκονται στην υλοποίηση του Horizon 2020 και επομένως η σταθερότητα και η αλλαγή είναι σημαντικά με την έννοια ότι η υποδομή είναι ιδιαίτερος δαπανηρή και επίσης υπάρχει και μία πολύ σημαντική ε, και ε, πολύτιμη γνώση ε, όσον αφορά το ίδιο το σύστημα, έτσι ώστε πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεκτικός σχετικά με τα αποτελέσματα τα οποία μπορούν ε, να, να, τα στοιχεία που μπορούν να τροποποιηθούν. Ε, και ε, βεβαίως εάν αλλάξει το σύστημα θα πρέπει να πληρωθούν και πολλά χρήματα όσον αφορά σε παροχή συμβουλών για την αντιμετώπιση του νέου προγράμματος. Δεύτερον, σε επίπεδο κρατών μελών, σε επίπεδο πανεπιστημίων, κέντρων έρευνας, μικρομεσαίων επιχειρήσεων μπορεί να προκύψουν διαφορετικές εφαρμογές των ε, αλλαγών. Και βεβαίως δεν μπορεί να υπάρξει όμως καμία διαφοροποίηση όσον αφορά την υλοποίηση και την ερμηνεία των ε, νομικών, ε, ε, των κανόνων γενικά, διότι είναι απαραίτητη και η νομική σαφήνεια και ασφάλεια όσον αφορά το πρόγραμμα αυτό. Και οπωσδήποτε ε, οπωσδήποτε ο δικαιούχος περιμένει στο τέλος να πάρει τα χρήματά του πίσω. Το τρίτο δίλημα είναι τα συμφέροντα των δικαιούχων και τα συμφέροντα της Ευρώπης. Αυτό συνδέεται με την επιλογή των συστημάτων επιστροφής των χρημάτων, με την έννοια ότι αυτή η επιστροφή προϋποθέτει την κάλυψη ε, την πλήρη κάλυψη του κόστους ε, των ε, δικαιούχων, ενώ ενδεχομένως το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήταν να προχωρήσει με καταποκοπήν αποζημιώσεις. Ένα άλλο δίλημα, το οποίο είναι και πάρα πολύ ε, ευαίσθητο αν θέλετε που αφορά την αριστεία και την ε, περιφερειακή γεωγραφική εξάπλωση. Πώς είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη είναι οι διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης που όλες συμμετέχουν ε, στο πρόγραμμα και μάλιστα ο χάρτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ότι δεν είναι ισομερής η γεωγραφική κατανομή στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα προκύπτει προβληματισμός σχετικά με την ε, ισορροπία που πρέπει να υπάρχει όσον αφορά την ε, ε, όσον αφορά την ισορροπία και την, την ίση κατανομή των κονδυλίων. Ένα πέμπτο και τελευταίο δίλημα αφορά την λογοδοσία και την ιδιοκτησία ε, εδώ μπορούμε να προχωρήσουμε προς ε, την κατεύθυνση της, ε, της αυτοδιαχείρισης, self-management των δικαιούχων, αλλά βεβαίως χωρίς να λησμονούμε τη λογοδοσία την οποία οφείλουν και οι δικαιούχοι, αλλά και η πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνει τα χρήματα. Το τελευταίο μου κεφάλαιο θα αφορά τις προτάσεις μας, ε, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τις παρατηρήσεις που κάναμε ε, στοιχείων και θεμάτων που σχετίζονται με την ε, υλοποίηση του προγράμματος Horizon 2020. Ένα θέμα είναι αρκετά απλό αλλά και δύσκολο να επιτευχθεί δηλαδή μια λογική χρονική διάρκεια ανάμεσα στην έγκριση και το, την υλοποίηση των ε, νομικών πράξεων η Κομισιόν αλλά και οι δικαιούχοι θα πρέπει να υλοποιήσουν ένα σύστημα εν τέλει από τη μία μέρα στην άλλη γιατί δεν έχουν πλέον πολύ ε, χρόνο στην διάθεσή τους και επομένως γίνεται πιο περίπλοκη και πιο δύσκολη η σωστή υλοποίηση ενός τέτοιου περίπλοκου προγράμματος. Επίσης, θα πρέπει να αξιολογηθεί η περαιτέρω χρήση απλουστευμένων, ε, απλουστευμένων επιλογών εναλλακτικών όσον αφορά το κόστος και ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν εργαλεία όπως είναι ε, ή είναι καταβολή ε, ή τα ε, βραβεία. Και βεβαίως και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να είναι σταδιακή η υλοποίηση η Κομισιόν ξέρει πώς να αντιμετωπίζει απλουστευμένες διαδικασίες κόστους και ξέρει και περίπου πώς η δικαιούχοι μπορεί να αντιδράσουν ε, σε μια απλουστευμένη διαδικασία επιστροφής ε, εξόδων. Επίσης, ε, διαπιστώσαμε ότι όσον αφορά τον οικονομικό έλεγχο, εάν υπάρχουν guidelines, κατευθυντήριες γραμμές ή παραδείγματα, ε, ε, θεωρούνται ε, ως μη δεσμευτικοί κανόνες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο οικονομικός έλεγχος, το audit όλων των στρωμάτων να παρέχει προ να παρέχει κάποιες προτάσεις και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που δεν θα είναι δεσμευτικές. Επίσης, θα πρέπει να δεχτούμε κατά κάποιο τρόπο όσον αφορά την αποδοχή μάλλον ε, των πρακτικών ε, ε, λογιστικών πρακτικών των δικαιούχων. Εδώ υπάρχουν κάποια ζητήματα. Βλέπουμε ότι σε μεγάλες εταιρείες μπορούν τα λογιστικά τμήματα να συμμετέχουν στο ορίζον 2020, αλλά ε, ε, ενδεχομένως μπορεί να δημιουργήσουν και ένα δεύτερο πιο μυστικό λογιστικό ε, σύστημα έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις περιπλοκότητες του, του συστήματος ενώ δεν έχουν την ίδια, τις ίδιες δυνατότητες κάποια ερευνητικά κέντρα ή ενδεχομένως κάποιες, κάποιοι δήμοι κλπ. Θα πρέπει να αποφευθεί ε, αυτή η λογιστική διαφοροποίηση, καθώς επίσης και η, ερμηνεία, η διαφορετική ερμηνεία των κανόνων από περιφέρεια σε περιφέρεια. Επίσης, θα πρέπει να αναγνωριστούν οι καλές προτάσεις προγραμμάτων ε, στον ορίζοντα 2020 και σε άλλα προγράμματα μέσα από μια προσέγγιση one-stop shop. Ε, είδαμε ότι πολλοί ε, υποψήφοι ε, τελικά απογοητεύονται από την διαδικασία, ενώ το πρόγραμμά τους ήταν ε, καλής ποιότητος. Και εδώ βεβαίως μία προκύπτει το πιο προκλητικό ας πούμε ερώτημα. Δεν είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε ε, δεν μπορεί να δούμε τα προγράμματα ξέχωρα το ένα από το άλλο. Ίσως θα πρέπει να δημιουργήσουμε μία δομή όπου τα διάφορα σιλό ε, συνδυάζονται ε, μεταξύ τους. Γιατί τα χρήματα είναι πολλά και η δουλειά είναι πολύ. Νομίζω ότι σας έδωσα αρκετές πληροφορίες με αυτή την σύντομη μικρή μου εισαγωγή. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια τώρα. Ευχαριστώ. Αξιότιμη Πρόεδρε. Ε, εκπρόσωποι του Ελεκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση αυτή από το Ελεκτικό Συνέδριο, για την απλούστευση των προγραμμάτων πλαίσιο των ερευνητικών από τότε που έφτασα στο Κοινοβούλιο πριν από τέσσερα χρόνια, ζητούμε απλούστευση της χρηματοδότησης και του κοινοτικού δικαίου γενικά. Δεν είναι εύκολο αυτό το εγχείρημα. Θα πρέπει όμως η Δημοσιονομική Αρχή να βρει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην εμπιστοσύνη και στον έλεγχο. Τι εννοώ με αυτό. Ε, ε, πολύ εύκολα το περιγράφουν τα διλήμματα που μας αναφέρεται, Παράδειγμα, ορίζον 2020, που είναι πάρα πολύ περίπλοκο εγχείρημα λόγω των διαδικασιών, ε, των κανονισμών, των κατευθυρίων γραμμών και πολλαπλά χρηματοδοτικά μέσα. Όλα αυτά επιφέρουν ένα κίνδυνο αναποτελεσματικότητας και παρατυπιών, ακριβώς επειδή είναι τόσο περίπλοκο. Και χαίρομαι που σε ένα τέτοιο ε, πρόγραμμα χρησιμοποιείται πιλωτικά για να δούμε ε, καταποκοπή ποσά για έμεσο κόστος, για κάλυψη κάποιων δαπανών κτλ. Έστω και πιλωτικά. Και με βάση τα όσα έχει αναλύσει το ελεκτικό συνέδριο για την έρευνα, τα καταποκοπή ποσά θα μπορούσε να είναι ένα μοντέλο ε, που να προσφέρεται. Δίνει μια σχετική απλοποίηση ιδιαίτερα όταν συμμετέχουν νέοι ερευνητές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ε, νέοι ε, ε, εταίροι στο πρόγραμμα αυτό το ερευνητικό. Υπάρχουν και κριτήρια επιδόσεων που εξασφαλίζουν την προστιθέμενη αξία. Δεν θα πρέπει να ανησυχεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εδώ δεν μιλώ μόνο για το πρόγραμμα πλαίσιο, το ένατο τώρα το ερευνητικό, αλλά και την επόμενη περίοδο. Είναι ενθαρρυντικά λοιπόν αυτά ε, για τους συμμετέχοντες, γιατί ε, η προσοχή τους θα πρέπει να εστιάζεται στην ίδια την έρευνα και όχι στη διαχείριση του ερευνητικού προγράμματος. Οι ερευνητές θα πρέπει να ε, ασχολούνται με την ουσία του προγράμματος και όχι με την κάλυψη γραφειοκρατικών ε, υποχρεώσεων και διοικητικών. Σας ευχαριστώ για τη συστάση και την πρότασή σας στο ελεκτικό συνέδριο. Συμφωνώ απολύτως με όλα όσα είπατε και περιμένω και ε, για τον ορίζοντα 2020 τη δημοσίευσή σας το 2018. περιμένω να ακούσω τι θα πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απλούστευση. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Ο κύριος Σχετχόφσκι ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω κάτι σε σχέση με τα όσα είπε προηγουμένως η Μαρτίνα, αλλά να τα πω τσεχικά καλύτερα, γιατί νομίζω ότι εκφράζομαι καλύτερα στη μητρική μου γλώσσα και θα, θα σας φάω και τόσο χρόνο όσο αν τα έλεγα στα αγγλικά. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, το ε, Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση σας για την ενδεχόμενη απλούστευση ε, των ερευνητικών προγραμμάτων πλαίσιο. Θέλω να ευχαριστήσω και τη Μαρτίνα που ανέφερε τα βασικότερα προβλήματα στο κείμενό της. Αυτά τα προβλήματα τα αντιμετωπίζουμε χρόνια ολόκληρα. Ακούσαμε ότι τέσσερα χρόνια περιμένουμε μία μεταρρύθμιση που δεν έρχεται ποτέ. Τα ίδια έλεγα ε, προηγουμένως για την έκθεση Κάντεμπαχ ακριβώς. Υπάρχει χώρος για πλούστευση βέβαια. Δεν χωράει καμία αμφιβολία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περίπλοκες δομές στα προγράμματά της και είναι ένα γραφειοκρατικό τέρας που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες και στις εξελίξεις και στα θέματα που απασχολούν την ερευνητική κοινότητα. Όπως ακούσαμε από τον κύριο Βιώτη, που είναι εισηγητής για τον προπολογισμό του 2019, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αυτές τις τεράστιες προκλήσεις. Η βιομηχανία μας δεν είναι ανταγωνιστική, χρειάζεται να τονωθεί. Όταν ε, συζητούμε σήμερα για το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα, ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα ε, προγράμματα ε, και οι διαχειριστές τους ε, τρομάζουν μπροστά σε αυτή τη γραφειοκρατία που τους αποτρέπει και τους αποθαρρύνει να προχωρήσουν σε ε, αιτήσει για χρηματοδότηση. Και αυτό οδηγεί σε γεωγραφικές ανισορροπίες. Κοιτάξτε πόσες χώρες από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα. Είναι σαφέστατη έλλειψη ισορροπίας και πολύ εύκολα μπορεί κανείς να την ανοιχνεύσει. τα ευρωπαικα κρατη κράτη-μέλη που έχουν ε, συνηθίσει να συμμετέχουν σε αυτά τα ερευνητικά προγράμματα πλέον εκτούν. Ας σταματήσουμε αυτή τη γραφειοκρατική υπανάπτυξη και αυτό το λαβύριθο. Ας ανοίξουμε τις πόρτες σε καινοτόμα προϊόντα και ιδέες. Συμφωνώ με το ελεκτικό συνέδριο σε ό,τι αφορά την απλούστευση ε, των πληρωμών, ιδιαίτερα σε πρώιμα στάδια, ε, που είναι πάρα πολύ κρίσιμες για μικρές εταιρείες και μικρά προγράμματα που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ε, την τεράστια αυτή συγχρηματοδότηση. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει να μας αναφέρει επιτυχίες στο συγκεκριμένο τομέα ελπίζω να αξιοποιήσουμε και τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, ιδιαίτερα της ψηφιακής τεχνολογίας, για την ε, διεκπαιρέωση των αιτήσεων για ε, τη λογιστική επίσης διεκπαιρέωση. Ε, χαίρομαι και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη συγχαίρω για την ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει και για άλλες ενέργειες της. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εκπαιδεύει ειδικευμένο προσωπικό στα κράτη-μέλη για να βοηθούν την υποβολή των αιτήσεων τους ενδιαφερομένους. Να τους βοηθήσουν να περάσουν αυτόν τον ε, γραφειοκρατικό λαβύρινθο, να έχουμε ενεργή και όχι παθητική παροχή συμβουλών και όχι χιλιάδες σελίδες θολές και ε, δυσνόητες κατευθυντήριες γραμμές που χωράνε και πάρα πολλές ερμηνείες ανάλογα με το κράτος μέλος. Τόσο συχνά ακούμε από τα διάφορα κράτη-μέλη ότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να ερμηνευθούν κατά το δοκούν και οι αρμόδιες ελεκτικές αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιλέξουν την ερμηνεία που τους βολεύει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να τα εγκρίνει όλα αυτά γιατί είναι πάρα πολύ ε, θολές και συγκεχημένες οι κατευθυντήριες γραμμές. Θέλω να ακούσω λοιπόν τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι προτίθεται να κάνει για να απλουστεύσει τη χρηματοδότηση στην έρευνα και την ανάπτυξη. Και με χαρά περιμένω και την επόμενη ειδική έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you very much, Chair. Mr. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Ευχαριστώ πολύ τον ε, κύριο Μπρένικ Μάιερ και τους βουλευτές. Πρέπει να πω ότι εκτιμούμε αυτό το σημείο για την απλούστευση και θέλω να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο. Γιατί το εκτιμούμε, διότι είναι επίκαιρε οι συμβουλές ε, σε να μην υποτίθεται ότι θα έχουμε τις νέες προτάσεις ε, για το προσεχές πρόγραμμα πλαίσιο. Εκτιμούμε όμως τις συμβουλές και για έναν ακόμη λόγο. Δείχνουν ε, τα διλήμματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο τομέα της απλούστευσης και αντικατοπτρίζουν και την εμπειρία μας ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο πολύπλοκο από την απλούστευση. Άρα συμφωνούμε απόλυτα με την έννοια αυτή που δίνει στο θέμα το ελεκτικό συνέδριο. Παρά τώρα το γεγονός ότι είναι πολύπλοκη απλούστευση, έχουμε πετύχει πολλά, υπάρχει η ευρεία συμφωνία. ως προς το Τεωρίζον 2020 έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο στον τομέα της απλούστευσης και αποτελεί ένα ορόσημο. Αυτή την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου θα διαβάσετε ότι αναφέρεται στην ευρεία χρήση επιλογών απλουστευμένου κόστους δημιουργία κοινού κέντρου στήριξης, participant board κτλ. Άρα έχουμε πρόοδο και αυτό αναγνωρίζεται από τους διάφορους ενδιαφερομένους και Βέβαια, θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Πρέπει να σημειώσουμε ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο. Οι συμβουλές λοιπόν του ελεγκτικού συνεδρίου είναι πολύτιμες. Εν συντομία τώρα θα ήθελα να σχολιάσω αυτά τα οποία αναφέρει στην έκθεσή του το ελεκτικό συνέδριο για το χρονοδιάγραμμα ε, μεταξύ έγκρισης και εφαρμογή των νομικών πράξεων. Αυτό είναι μια πρόκληση γενικώ για τους ε, συνομοθέτες κομισιών. Θα προτείνει κανόνα 30 μήνες πριν από την έναρξη ισχύω. Η διαδικασία συναπόφασης όμως θα πρέπει να επιτέει να συνεισφέρει στην γρήγορη εφαρμογή. Όταν προτείνουμε το νέο νομικό πλαίσιο, θα επεξεργαστούμε, με τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς και το θέμα των εκτελεστικών πράξεων. Να γνωρίζουν δηλαδή από την αρχή πώς σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε τους κανόνες ενδιαφερόμενοι. Δεύτερον, αξιολόγηση περαιτέρω χρήσης ε, των ε, επιλογών απλουστευμένου κόστους ε, κάποια καταποκόπη ποσά λοιπά. Στον ορίζοντα 2020 το 30 περίπου των δαπανών γίνεται ακριβώς με επιλογές τέτοιες, απλουστευμένου κόστους. Για το έμεσο έχουμε την Μαρσιλοτόσκα Κιουρί, το βραβείο το μέσο για τις μικρές επιχειρήσεις, άλλα βραβεία και ξεκινήσαμε πρόσφατα πιλωτικά προγράμματα με καταποκοπή χρηματοδότηση, έναν διαγωνισμό στον νομιμέα της υγείας, έναν στην τεχνολογία και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας. Εκεί θέλουμε να έχουμε για την απόδειξη κάποιων κόνσεπτ, επίσης ε, καταποκοπή διαδικασίες και για το shift to rail. Γιατί έχουμε θεσπίσει τα μέτρα αυτά ακριβώ γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι μπορούν να οδηγήσουν σε απλούστευση και να μειώσουν τα ποσοστά σφάλματος. Όμως, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προκλήσεις και διλήμματα σε ό,τι αφορά τη θέσπιση των καταποκοπήν ποσών και σημείωσα πολύ προσεκτικά την παρατήρηση του κ. Μπρένικ Μάγερ ότι πρέπει να γίνει βαθμιαία αυτό και Το ίδιο πιστεύουμε και εμείς. Η θέσπιση καταρχάς κατά αποκοπήν ποσών ε, γύρει ζητήματα. Καταρχάς στο επίπεδο των εμπλεκομένων φορέων, των δικαιούχων. Γιατί? Διότι για δεκαετίες οι δημόσιες αρχές, πανεπιστήμια, ερευνητικοί οργανισμοί, ήθελαν ε, την αναφορά από το πραγματικού κόστους ώστε τα πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα να μπορούν πραγματικά να δείξουν στις δημόσιες αρχές το κόστος της έρευνας. Πραγματικά κάναμε αγώνα να έχουν συστήματα κόστος που θα αντικατοπτρίζουν το κόστος έρευνας. Τώρα, υπάρχει φόβος ότι θα μειωθεί η χρηματοδότηση λόγω αυτών των καταποκομικών ποσών και τρίτον, το είπε και ο κύριος Μπρένικ Μάιο νομίζω, Αυτά τα καταποκοπήν ποσά απαιτούν αλλαγή διοικητικών και δημοσιονομικών πρακτικών και γύρονται και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ευθύνη των εταίρων σε ερευνητικά προγράμματα. Άρα θέλουν να δουν οι εμπλεκόμενοι φορείς πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα ποσά. Δεν είναι όμως 100% πώς να το πω, θετική και θετικά διακείμενη σε κάτι τέτοιο. Η εισαγωγή των καταποκοπήν ποσών και, ε, θέτει και ζητήματα λογοδοσίας. Πρέπει εκ των προτέρων να αξιολογήσουμε πολύ προσεκτικά το ενδεχόμενο κόστος των ερευνητικών προγραμμάτων. Και αυτό απαιτεί μια πολύ διαφορετική προσέγγιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των ερευνητικών προγραμμάτων. Ε, σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση, την παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών, στοιχεία δηλαδή που άπτονται της λογοδοσίας για τα καταποκοπήν ποσά. Παρά τα αυτά, εμείς είμαστε έτοιμοι στο επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο, κατά περίπτωση να θεσπίσουμε περαιτέρω καταποκοπήν ποσά, όπου κρυθεί σκόπιμο κάτι τέτοιο. Τρίτο σημείο συμφωνούμε σε ό,τι αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές, ότι πρέπει να βοηθούν τους συμμετέχοντες και να μην θεωρούνται δεσμευτικές. Και σίγουρα θα ακολουθήσουμε τη σύσταση αυτή. Σε ό,τι αφορά την ευθυγράμμιση των λογιστικών πρακτικών των δικαιούχων, αυτό το ζήτημα έχουμε χρόνια που το αντιμετωπίζουμε. Η πρόκληση σε ό,τι αφορά την αναγνώριση των λογιστικών πρακτικών των συμμετεχόντων και των δικαιούχων το εξή. Ο δημοσιονομικός κανονισμός ξεκάθαρα θεσπίζει τους κανόνες, προβλέπει κανόνες σαφείς για το επιλέξιμο κόστος. Σε εθνικό επίπεδο όμως ή σε επίπεδο δικαιούχων υπάρχουν κάποιες πρακτικές ε, λογιστικής καταγραφής του κόστους που δεν επιτρέπουν να καταγραφεί αυτό το κόστος που εμείς θεωρούμε ότι είναι επιλέξιμο. Εξού και είναι δύσκολο εμείς να δεχθούμε τις λογιστικές αυτές πρακτικές. Καθότι συχνά δεν επιτρέπουν τον επανυπολογισμό του κόστους ενός προγράμματος. Πολλά πανεπιστήμια, ερευνητικοί οργανισμοί αλλά και επιχειρήσεις έχουν κάποια cost center που όμως δεν ε, εντοπίζουν το κόστος ενός συγκεκριμένου προγράμματος. Γι' αυτό λοιπόν θα το μελετήσουμε περαιτέρω το θέμα για να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να δεχθούμε τις λογιστικές πρακτικές των συμμετεχόντων και των κρατών μελών. Αλλά είναι σημαντικό αυτά, ε, αυτές οι πρακτικές να συνάδουν με τους περιορισμούς δημοσιονομικού ανισμού. Τέλος, η μοναπευθυντική θηρίδα, το one-stop shop για τη χρηματοδότηση. Όπως επισημαίνει το ελεγκτικό συνέδριο, στον ορίζοντα 2020 μόνο είχαμε πάρα πολλά προγράμματα, αλλά το 14 μόνο 100 χρηματοδοτήθηκε. Επειδή πολλά προγράμματα, αν και είναι εξαιρετικά, είναι πάνω από το κατόφλι. Εξού και έχουμε το φλό αριστείας. Μπορεί να υπάρξει μεταδότηση από τους εθνικούς προπολογισμού ή από τα διαρκτικά ταμεία. Πιστεύουμε ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα ταμεία αυτά για να χρηματοδοτήσουν και αυτά τα προγράμματα, αυτά τα έργα που θεωρούνται άριστα, έργα αριστεία. Τι συμφορήσεις υπάρχουν όμως ότι δεν δέχονται οι χρηματοδότες τα προγράμματα που έχουν εξελιχθεί στο νωρίς το 2020 να λάβουν χρηματοδότηση από τα εθνικά συστήματα χρηματοδότησης ή μέσω των διαθερωτικών ταμείων. Στις προσεχείς δημοσιονομικές προοπτικές θα φροντίσουμε να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση για τέτοια έργα να είναι μια επιλέξιμη δράση στο πλαίσιο των ευρωτικών ταμείων. Δεύτερη συμφόρηση. Αν γίνει δεκτό ένα έργο στο νόριο του 2020, ένα project, ας πούμε, μιας ΜΜΕ, το ποσοστό είναι 120% για την χρηματοδότηση. Και οι κανόνες πεκρατικών ενισχύσεων δεν εφαρμόζονται, δεν ισχύουν. Αν θέλουν τα κράτη-μέλη να χρηματοδοτήσουν τέτοια έργα στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων χρηματοδότησης ή στο πλαίσιο των διαθροτικών ταμείων, των προγραμμάτων για το διαθετικό ταμείο, υπάρχουν διαφορετικοί κανόνε για την επιλεξιμότητα του κόστου. Και αυτό κυρίω λόγω των κανόνων περικρατικών ενισχύσεων. Έχουμε πολύ στενέ επαφέ, ε, είμαστε σε επικοινωνία με του συναδρόμου από τη ΓΑΜΑ Ανταγωνισμού και έχουμε καταλήξει σε συμφωνία. όταν έχουμε προγράμματα επιλέξιμα για τον ΙΟΣΤΟ 2000 που έχουν το σήμα αριστεία, θα πρέπει στο μέλλον να μπορούν να, χρησιμο... να χρηματοδοτηθούν με βάση τους ίδιους ακριβούς κανόνες που ισχύουν για τον ορίζοντα 2020. Αυτά λοιπόν ως δική μας ανταπόκριση στο πέμπτο, ε, στην πέμπτη πρόταση του ελεκτικού συνεδρίου. Είμαστε πεπισμένοι ότι έχει γίνει μεγάλη πρόοδο στο ορίζοντα 2020 και είμαστε και αισιόδοξοι ότι θα μειωθούν και τα ποσοστά ασφάλματος. Βέβαια, απαιτείται περαιτέρω πρόοδο στο μέτωπο τη απλούστευσης και κατά περίπτωση ε, θα δοκιμάσουμε το κατά πόσο είναι ενδεδειγμένη η αυξημένη χρήση των ε, προσταυμένων επιλογών κόστους και θα δούμε και πόσο μπορούμε να δεχθούμε τις λογιστικές πρακτικές των δικαιούχων εφόσον συνάδουν με τις δημοσιονομικούς κανονισμούς. Ευχαριστώ. Ε, ο πολύ συνάδελφος Τσέλερ ξαναζήτησε το λόγο. Όχι, εντάξει, έχει καλυφθεί. Ωραία αναφερθήκατε στο δημοσιονομικό κανονισμό και ανησυχώ γιατί αυτά που μας είπατε διαφέρει κατά πολύ ε, από εκείνα που μας είπε και μας έδωσε στο δημοσιονομικό κανονισμό η Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού για τις συνήθεις λογιστικές πρακτικές που θα πρέπει να ισχύουν και θα πρέπει να υπάρχουν και απαγορεύσεις ελέγχου για το διατάκτη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάποιους τομείς. Και μετά από όσα μας είπατε τώρα, εγώ το βρίσκω αυτά τραγικά. Δεν συνάδουν. Μήπως να το συζητήσετε με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Πράγματα που είναι ασυμβίβαστα μεταξύ του θα πρέπει να είναι ασυμβίβαστα και να αναγνωρίζεται. Και όποιος θέλει λεφτά από την Ευρώπη θα πρέπει να υποκλίνεται και να τηρεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Τι να κάνουμε τώρα, λυπάμαι πάρα πολύ να σας ρωτήσω, στο νέο δημοσιονομικό κανονισμό ποιες ε, είναι οι επιπτώσεις για σας, ε, βλέπετε περιορισμούς για τη δουλειά σας. Ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός είναι κάτι που θεωρούμε ιδιαίτερα θετικό. Γιατί σε εμά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας δίνει την απαραίτητη ευελιξία ε, από πολλές πλευρές. Καταρχάς, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι στήριξης ε, ο δημοσιονομικός κανονισμός προβλέπει ε, την επιστροφή των πραγματικών εξόδων αλλά ε, και πολλές άλλες δυνατότητες επιστροφής δαπανών επιτρέπονται. Και ιδιαίτερα σημειώνουμε ότι έχουμε νέες κατηγορίες για την επιστροφή δαπανών που βασίζονται σε επιδόσεις ή προσανατολίζονται στις επιδόσεις και αυτό είναι σίγουρα ένας τομέας που θα ελέγξουμε και από εκεί και πέρα λοιπόν στόχος μας ποιος είναι ε, στους κανόνες συμμετοχής μας να προσαρμοστούμε όσο γίνεται με τους κανόνες του δημοσιονομικού κανονισμού για να έχουμε ενιαίους κανόνες και για την έρευνα και για την καινοτομία. Ενιαίοι κανόνες είναι κάτι για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Και μόνο όταν έχει ενιαίου κανόνε είναι ουσιαστική απλούστευση, γιατί χάνονται οι αντιφάσει και, και ε, εκτοπίζονται. Λοιπόν, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι τα συστήματα τήρησης λογιστικής καταγραφής τα βιβλία. Σε σχέση με τα όσα είπατε, πώς βλέπετε αυτό που λέει ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός, ότι εν μέρη υπάρχει ένα ασυμβίβαστο ε, στο διαχωρισμό των δαπανών στα κράτη-μέλη, ενώ εσείς το χρειάζεστε αυτό. Κοιτάξτε, για την έρευνα και την καινοτομία είναι βασικό το εξής. Να εργαζόμαστε σε συστήματα όπου ε, το δαπανηθέν ε, κόστος να επιστρέφεται και τα εθνικά συστήματα θα πρέπει να μας δίνουν τη δυνατότητα, να δίνουν τη δυνατότητα να ταυτοποιείται το κόστος, οι δαπάνες που έχουν πραγματικά ε, καταβληθεί. Υπάρχουν εθνικά λογιστικά συστήματα που δεν είναι προσανατολισμένα σε αυτό. Δηλαδή, να καταγράφει σε κάθε έργο το μεμονωμένο κόστος και να μπορεί κανείς να ε, το εντοπίσει. Σε πολλές εταιρείες και σε πολλά πανεπιστήμια υπάρχουν ε, τέτοια κέντρα υπολογισμού του κόστους που υπολογίζουν μόνο το κόστος εργασίας. Ε, για το Ινστιτούτο. Αλλά με βάση αυτή τη λογιστική και αυτά τα βιβλία είναι δύσκολο να διαπιστώσεις πόσες είναι οι παραγωγικές ώρες που έχει αφιερώσει ένας ερευνητής σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα. Και μας ε, όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι γνώμον το πραγματικό κόστος. Αν δεν μπορεί ένα λογιστικό σύστημα να το πιστοποιήσει αυτό, τότε μας δυσκολεύει πάρα πολύ εμάς να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό απολύτως. Ευχαριστώ πολύ. Επιθυμεί το λόγο το ελεκτικό συνέδριο ξανά. Ευχαριστώ κυρία Γκρέσλε. Πάρα πολύ σύντομα. Θα σας τα πω. Ε, Ο ρόλος ε, του ελεγκτικού συνεδρίου είναι πάρα πολύ μικρός με την έννοια ότι εμείς ε, κάνουμε σε αιτήσια βάση αναλύσεις και τις κάνουμε και τις ειδικές μας εκθέσεις στις οποίες ε, υποβάλλουμε σειρά προτάσεων ε, στο, στους νομοθέτες και στην πλευρά της Κομισιόν. Ε, και εμείς υποβάλλουμε τις προτάσεις που θεωρούμε λογικές και βεβαίως είμαστε πάντα στη διάθεση όλων έτσι ώστε να μελετήσουμε την αποτελεσματικότητα τέτοιων προγραμμάτων και βεβαίως να υποβάλουμε και ε, προτάσεις ε, προς ε, τους νομοθέτες έτσι ώστε να κάνουν τη σωστή νομοθεσία. Ευχαριστούμε. Δεν μπορούμε παρά να σας ενθαρρύνουμε. Γιατί είδαμε ότι στο πρόγραμμα εργασίας σας στο ελεκτικού συνεδρίου φέτος δεν αναφέρεται πουθενά η έρευνα. Έχετε άλλες προτεραιότητες. Καλό θα ήταν κάποια στιγμή να μας κάνετε ειδική έκθεση ακριβώς για την έρευνα. Ναι, πέρα από την ετήσια έκθεσή μας και τη δήλωση αξιοπιστίας και για τον ορίζοντα 2020, κάνουμε και έλεγχο λογιστικό επιδόσεων του ορίζοντα 2020 βάσει μιας μελέτης έρευνας για τους δικαιούχους του προγράμματος αυτού και σε εργαστή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσπαθήσουμε να εκπονήσουμε και χρήσιμες εκθέσεις και προτάσεις για την εκτέλεση του Οριζόντα 2020 στο τρέχον πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ. Εξαντλήσαμε την σημερινή μας ημερήσια διάταξη, οπότε είναι η επόμενη συνεδρία στις 14 Μαΐου. Καλά να περάσετε και καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.